Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται αυτή τη στιγμή έχουν μόνο 2.888 και κάτι τετραγωνικά μέτρα. Είναι πολύ δύσκολο για αυτές τις ε, ε, ε, συμπράξεις κατά κάποιο τρόπο να στεγαστούν σε ένα τόσο μικρό χώρο. Θα είναι χρήσιμο λοιπόν να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, να έχουμε ένα νέο ε, χώρο και να αποφύγουμε αυτό το οποίο γίνεται τώρα, να έχουμε τέσσερα άτομα στο ίδιο γραφείο, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ποια είναι τα προβλήματα και η, η πρόθεσή μας είναι να έχουμε ένα κτίριο στο, στην Τουαζόν Ντό στις Βρυξέλλες. Έχουμε λοιπόν καλές συνδέσεις ε, σε επίπεδο συγκοινωνιών. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να υπάρξει αυτή η ανακαίνιση του κτηρίου για να προσαρμοστεί στις ανάγκες μας και επίσης δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Ε, το κτίριο δεν είναι μονάχα ελεύθερο αμοιάντου αλλά έχει πιστοποιηθεί ότι είναι απόλυτα ασφαλές ως προς τους κινδύνους ύπαρξης ε, ασβεστίου. Έχουμε ένα, προβλέπεται να υπάρχει ένα συμβόλαιο 15 ε, ετών με δυνατότητα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 να διακοπεί αυτό το Συμβούλιο, γιατί τότε θα πρέπει να είναι η στιγμή που θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για το, για το κατά πόσο θα συνεχιστούν αυτά τα πέντε προγράμματα, οι κοινέ συμπράξει αυτού του είδου. Με την παρουσία <clears throat> βέβαια όλων των ε, ομάδων των πέντε αυτών προγραμμάτων στο ίδιο κτίριο. Θα έχουμε εξοικονομήσεις γιατί μπορούμε να εξοικονομήσουμε παραγωγικά υπηρεσίε ασφαλείας ή καθαρισμού κτλ. Μπορούμε να έχουμε επομένω και αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και θα έχουμε περίπου 4.200 τετραγωνικά μέτρα ε, επιφάνεια γραφείων και είναι 175 ε, ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η, το μίστομα για τις πέντε κοινές αυτές επιχειρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πραγματικά μικρό το τίμημα το οποίο ε, θα έχουμε στην περίπτωση αυτή για τα κτίρια αυτά και η επιλογή αυτή προς το παρόν φαίνεται ότι είναι η καλύτερη δυνατή θα μας κοστίσει 1,9 1,19 εκατομμύρια συνολικά για τα 7 χρόνια θα είναι 9.278 και κάτι ψηλά μέχρι το 2017. Υπήρξαν 27 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, περάσανε μία διαδικασία και έχουν μείνει μονάχα έξι υποψήφοι και αναφέρονται εδώ οι τρεις καλύτερες προτάσεις. Η διαδικασία αυτή έγινε με διαδικασία προσβολής προσφορών σε όλη την Ευρώπη και πιστεύω ότι γενικά το συνολικό κόστος θα καλυφθεί κατά 60% από τον ιδιωτικό τομέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μονάχα το 37%. Αυτό η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ως θετικό. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζω τι γίνεται με τις ε, υπηρεσίες αυτές τις αποκεντρωμένες, γιατί έχω μεγάλη πείρα για τα θέματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση αυτή δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα και εγώ επομένως μπορώ να υποστηρίξω αυτά τα οποία λέει η εισηγήτριά μας για την πολιτική κτίριων. dann haben wir das jetzt so miteinander beschlossen. Νομίζω ότι εάν δεν υπάρχει αντίρρηση έχει αποφασιστεί. Ωραία, μπορείς να διαδώσεις τις καλές ειδήσει για το θέμα αυτό, Μόνικα. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης και θα ξεκινήσουμε με τον εισηγητή μας και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να μας παρουσιάσει τη θέση του και μπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε συζήτηση. Ο Ιβάιλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ήδη το συζητήσαμε κάποιες φορές το θέμα που σας παρουσιάζω σήμερα ως έκθεση Uh, Η Επιτροπή μας θέλει να βοηθήσει το Κοινοβούλιο για την επέκταση, την παράταση της εντολής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την κάλυψη σημείων και δάνεια από εγγύηση για σχέδια. Λίγη τον Οκτώβριο του 2011. Θα πρέπει να φροντίσουμε να ολοκληρωθεί αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται έτσι να μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες της η τράπεζα. Για την ανανέωση της εντολής έχουμε πολύ συγκεκριμένο συμφέρον στο Κοινοβούλιο. Αφορά έξι επιτροπές για γνωμοδότηση Πολλές προτάσεις και ιδέες και σκέψεις κυκλοφορούν για την εξωτερική εντολή της τράπεζας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Κομισιόν για την άρεστη πρότασή της. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε σε συναπόφαση. Πρέπει να συμφωνήσουμε για το ίδιο κείμενο, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή βάση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την τράπεζα και πιο συγκεκριμένα τον πρόεδρο κύριο Μεστάντ για την διαθεσιμότητά της συνεχώς να συζητήσει όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτό μας διευκόλυνε στη δουλειά μας και θα βοηθήσει να διαμορφωθεί η τελική γνώμη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και τους οικειώδεις εισηγητές των άλλων ομάδων και τους συζητητές των άλλων πέντε επιτροπών. Θα σας παρουσιάσω σε γενικές γραμμές αυτό που προτείνουμε για την παράτηση της εξωτερικής εντολής. Πρώτο, Στόχος μας είναι να έχουμε περισσότερη συνοχή μεταξύ των δραστηριότητων της Τράπεζας και πολιτικών της Ένωσης. Και με την πρόταση εξασφαλίζουμε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας και των διαφόρων οργάνων της Ένωσης. Και με οριζόντιους στόχους και στόχους κατά περιφέρεια, κατά χώρα, έτσι ώστε η δραστηριότητα της Τράπεζας να συμπληρώνει τις δραστηριότητες και τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Δεύτερο, προτείνουμε να δοθεί με επιπλέον εγγύηση 2 δις ευρώ που ήταν στο αποθηματικό και να δώσουμε το δικαίωμα στην τράπεζα να χρησιμοποιήσει αυτή την εγγύηση για μετριασμό, προγράμματα μετριασμού της, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. Έτσι ώστε να βοηθηθεί μια από τις κύριες πολιτικές της Ένωσης που είναι η καταπολέμηση της, των επιπτώσεων της κλιματολογικής αλλαγής. Συζητήσαμε πολύ το ρόλο της τράπεζας σχετικά με τη δέσμευση της Ένωσης για στόχους ανάπτυξης, όπως τους ορίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι ιδέες ήταν πολλές και διεστάμενες. Δεν προτείνουμε την αλλαγή του προφίλ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι τράπεζα επενδύσεων και θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με τον επιτυχή τρόπο που λειτουργήσε ως τώρα. Ταυτόχρονα, επειδή πολλά από τα προγράμματα που ήδη τρέχουν έχουν επίπτωση στην ανάπτυξη, προτείνουμε τυπικά να δούμε ποια είναι η επίπτωση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων της ΕΤΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες. για να αξιολογήσουμε ακριβώς τι προσφέρουν οι δραστηριότητες της ΕΤΕ στην ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε πριν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα η ΕΤΕ να μελετήσει πολύ προσεκτικά το κάθε θέμα και ιδιαίτερα κάτω από το πρίσμα της ανάπτυξης της συγκεκριμένη χώρας. Να δώσει στοιχεία μετά του τι πέτυχε για την ανάπτυξη στην ε, χώρα που έλαβε τη βοήθεια Η τράπεζα έχει πει σαφώς προς το Συμβούλιο ότι χρειάζεται επιπλέον προσωπικό και περισσότερη πρόσβαση σε διάφορες άλλες επιδοτήσεις εκ μέρους της Ένωσης, ιδιαίτερα αν θέλουμε η ΕΤΕ να λειτουργεί σε λιγότερο αναπτυγμένε χώρες όπου δεν πληρούνται οι συνθήκες προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλος κίνδυνος των κεφαλαίων της τράπεζας. Προτείνουμε τυπικά καλύτερο συντονισμό μεταξύ της ΕΤΕ και των άλλων χρηματοδοτικών οργάνων. Είτε τράπεζες, είτε εθνικά ιδρύματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, αυτή η καλύτερη συνεργασία μας οδηγεί σε μελέτες που έγιναν μεταξύ επιδοτήσεων ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αφρική όπου η δουλειά γίνεται σε μια κοινή πλατφόρμα μεταξύ της ΕΤΕ και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Προτείνουμε να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η δραστηριότητα και να μελετήσουμε κατά πόσο αυτός ο μηχανισμός συνεργασίας όλων αυτών των φορέων μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Σας ειδοποιώ όταν το τέλος θα διαπραγματεύουμε το Συμβούλιο ένα από τα σοβαρά θέματα θα είναι οι οροφές. 26,8 δις ευρώ είναι η συνολική οροφή της τράπεζας. Κονδύλια κατά περιοχές. Η Ένωση ζήτησε από την ΕΤΕ τα τελευταία χρόνια να αυξήσει τη δραστηριότητά της σε μερικές και επιπλέον προσθέσαμε και χώρες επιλέξιμες που σημαίνει αν θέλουμε η τράπεζα να μείνει στις δραστηριότητες που έχει και πάλι θα χρειαστεί επιπλέον χρήματα. Εμείς προτείναμε αύξηση των οροφών η δημοσιονομική επίπτωση θα είναι μετά από δύο χρόνια περίπου 9%. νέα κονδύλια που θα πρέπει να προσθεθούν στο Ταμείο Εγγύσεων. Αυτό όμως θα έχει μόχλευση. Ψηλή μόχλευση το ποσό αυτό. Μέχρι και 15 φορές. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο της ΕΤΕ. Άλλο θέμα. το μέλλον της μελλοντικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της Ένωσης. Η εντολή που μελετάμε για την ΕΤΕΝ μέχρι το 2013. Με βάση την έκθεση που δόθηκε σε μια ομάδα σοφών υπό τον κύριο Καμτεσού, γνωστό εμπειρογνώμονα, πρότεινε διάφορες συγκεκριμένες λύσεις για να αυξηθεί η αποδοτική χρήση των κονδυλίων ανάπτυξης όπως ε, να δημιουργηθεί ενδεχομένως μια θεατρική εταιρεία της ΕΤΕ ενδιάμεσα κλπ. κλπ. Εμείς δεν μπορούμε να προδικάσουμε που θα οδηγήσει αυτή η συζήτηση. Πάντως επιβάλλεται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συζητήσουν το πώς τα διάφορα κονδύλια, ταμεία της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για την ανάπτυξη. Και να γίνει και μια ομάδα εργασία που να συζητήσει το θέμα αυτό και να καταλήξει σε ένα πόρισμα πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τη νέα εντολή μετά το 2013. Τέλος. Διαφάνεια περισσότερη δημόσια πληροφόρηση εκ μέρου τη τράπεζα, Πιο καλά διορθωμένη πληροφόρηση που δίνεται στο Κοινοβούλιο. Αξιολόγηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ένωση. Όλα αυτά θα τα δείτε υπάρχουν στην έκθεση. ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια πλήρη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να στηριχτούμε στις θετικές εμπειρίες της ΕΤΕ και να μην αφήσουμε να παρασφυρίσουν κίνδυνοι. Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν τελείωσε. Εμείς προτείνουμε και ένα χρονοδιάγραμμα 4 Νοεμβρίου για τροπολογίες στην έκθεση. Αν οι συνάδελφοι δεν έχουν αντιρρήσεις, προτείνω να το φέρουν πιο κοντά αυτή την ημερομηνία για να ψηφίσουμε την έκθεση τέλος Νοεμβρίου. γιατί ήδη το συζητήσαμε το θέμα και με συναδέλφους από άλλες επιτροπές συναντήθηκαν οι σκιώδει συγητές αν δεν υπάρχει αντίρρηση των συναδέλφων κύριε Πρόεδρε προτείνω να βάλουμε την ημερομηνία τροπολογικών 28 Οκτωβρίου για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρωτού αντιμετωπίσουμε άλλα θέματα, ίσως πρέπει να διευκρινίσουμε αυτό το, αυτό το σημείο. 28 Οκτωβρίου είναι η επόμενη Πέμπτη. Στις 12 η ώρα λοιπόν, αν συμφωνούμε όλοι, να είναι τότε η προθεσμία για την, ε, για την κατάσταση τροπολογιών, οπότε εγκαίρως μπορεί να γίνει η μετάφραση για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Νοέμβριο. Αν δεν βλέπω καμία, αν δεν υπάρξει κάποια Έχετε αντίρρηση. Μήπως μπορεί να είναι 29 Οκτωβρίου χωρίς αυτό να αλλάξει το χρονοδιάγραμμά σας. Απλώς αυτό ρωτώ. Αυτό θα ήταν πολύ βολικό για μένα. Και η 29η φαντάζομαι ότι θα είναι αποδεκτή. Εντάξει. Η νέα προθεσμία είναι 29 Οκτωβρίου στις 12. Την Παρασκευή λοιπόν που μας έρχεται στις 12. Σας παρακαλώ λοιπόν, όπως τόνισε ο κύριος ε, Κάλφιν, θα ήταν χρήσιμο, παρακαλώ, αν θέλω να απευθυνθώ στους δύο συντονιστές του ΕΛΚ. Σας λέω ότι σας παρακαλώ να δώσετε τη, λίγο περισσότερη προσοχή σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε ούτως ή άλλως τώρα και από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον οποίο δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που διαμορφώσατε και τις συνθήκες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ήρεμα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας, τον κύριο Κάλφιν, αλλά και τους εισηγητές των άλλων επιτροπών. Εμείς λάβαμε ένα σωρό ερωτήσεις. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτό σημαίνει πόσο πραγματικά εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία και οι εισηγητές και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου για το θέμα της ε, αναδιάθρωσης εντολής της ΕΤΕ. Να σταθώ τώρα στα διάφορα σημεία του εισηγητή σας. Πρώτο σημείο του κυρίου Κάλφιν. Να βελτιώσουμε την συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΕΤΕ και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ουσιαστικότατο σημείο αυτό. Οι εκτιμήσεις που γίνανε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κρίνουν ότι οι δράσεις της ΕΤΕ ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης, αλλά υπάρχει τρόπος να βελτιώσουμε αυτή τη συνέργεια και ζητιέται, και εμείς το προσυπογράφουμε αυτό, να υπάρχουν κοινοί προσανατολισμοί μεταξύ Κομισιών και ΕΤΕ για τις δράσεις της Ένωσης προς τα έξω. Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο. Διαπιστώνω λοιπόν όταν πηγαίνω στο εξωτερικό ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και η πιο σημαντική δηλαδή διότι άμα δούμε εμείς όλη την κοινή δράση κρατών, μελών και ένωσης είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές στον κόσμο. Χάνουμε όμως σε ορατότητα και σε δημοσιότητα διότι δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων πρωταγωνιστών αυτής της βοήθειας. Το προσυπογράφω λοιπόν αυτό που λέτε. Τώρα, η πρόταση, τα, τα δύο εκατομμύρια στην, της απόφασης του 2006 που είχαν μπει στο αποθεματικό να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των δράσεων κατά των κλιματικών αλλαγών. Φυσικά η ΕΤΕ προσυπογράφει αυτή την πρόταση διότι αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Τώρα αυτά τα δύο δις ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μία μόνη περιοχή του πλανήτη, πρέπει να βρούμε μία ισορροπία. Το Συμβούλιο πρέπει λοιπόν να αποφασίσει φυσικά θα δώσει συνέχεια σε αυτή την πρόταση. Τώρα το άλλο σημείο είναι ένα πιο λεπτό σημείο είναι πώς συμβάλλει η ΕΤΕ στους στόχους της χιλιετίας και κυρίως σε αυτόν τον πρωταρχικό στόχο που είναι η μείωση της φτώχειας. Ο εισηγητής σας λέει ότι δεν... Γιατί να μην αλλάξουμε το προφίλ της ΕΤΕ και να γίνει η ΕΤΕ να μια πραγματική τράπεζα επενδύσεων. Αν φυσικά εσείς το προτείνατε, το Συμβούλιο να ξέρετε θα το αρνιότανε, θα το απέρριπτε. Λέει ο εισηγητή σα όμως ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική η ΕΤΕ για τις επιπτώσεις των διαφόρων σχεδίων που χρηματοδοτεί στο περιβάλλον. Η οικονομική ανάπτυξη ελπίζουμε ότι θα έχει μία οικονομική μια θετική οικονομική επίπτωση και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Εμείς όμως δεν είμαστε εξοπλισμένοι να, στη χρηματοδότηση σχεδίων που καταπολεπούν άμεσα τη φτώχεια στην, για την παιδεία ή για την υγεία διότι αυτές, αυτά τα, αυτές οι πράξεις πρέπει να χρηματοδοτούνται με, με, με με προτιμησιακά επιτόκια και αυτό δεν μας το επιτρέπει το καταστατικό λειτουργίες μας. Θα πρέπει όμως η επίπτωση στην αναπτυξιακή διαδικασία να, να εκτιμάται με έναν καλύτερο τρόπο στις ε, συνδιαλλαγές μας εκτός Ένωσης. Αυτό γίνεται. Αλλά με δύο όρους που εσείς ο ίδιος αναφέρατε κύριε Σιγητά. Πρώτος όρος είναι να δεχθούμε ότι όντως μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό για τις ε, δράσεις μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας το λέω σαφέστατα το διοικητικό μου συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών όταν τους λέω να προσλάβουμε προσωπικό για ε, δουλειά στην ε, για δράσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το προσλάβουν αλλά όταν ζητώ να προσληφθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το προσωπικό έχω τρομερές αντιστάσεις πόσο μάλλον ε, και ακόμη μάλλον και οι χώρες οι οποίες έχουν δικές τους, ε, δικούς τους αναπτυξιακούς οργανισμούς εκτός ε, Ένωσης αρνούνται Συμφωνώ απόλυτα κύριε εισηγητά με, το, με αυτά που μας λέτε αλλά θα πρέπει να προσλάβουμε επιπλέον προσωπικό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ε, αναλύσεις των επιπτώσεων, να μπορούμε να έχουμε μία συνεχή παρακολούθηση των όλων δράσεων και δεύτερος όρος, το είπατε και εσείς ο ίδιο, να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη, μεγαλύτερη πρόσβαση σε προτιμησιακά επιτόκια. Διότι για να μπορέσουμε εμείς να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους ε, δράσεις ε, σε τρίτες ε, χώρες, σε φτωχές χώρες, πρέπει να έχουμε χαμηλά επιτόκια. Σήμερα εμείς δανείζουμε με επιτόκιο αγοράς. Για να έχουμε όμως εμείς προτιμησιακά επιτόκια, χρειαζόμαστε μία παρέμβαση εκ των έξω. Δηλαδή είτε τα κράτη-μέλη είτε τα μία εγγύσεων για να μπορέσουμε λοιπόν να χορηγούμε αυτά τα προτιμησιακά κονδύλια. Ένα τέταρτο σημείο που αναφέρατε κύριε Ισηγητά είναι η ανάγκη να βελτιώσουμε τον συντονισμό δύο μεγάλων οικονομικών οργανισμ, διεθνών οργανισμών Μα αυτό πάντοτε το επιμένω. Επιμένω πάντα σε αυτό. Η, τρα... η ΕΤΕ σήμερα προσκαλείται στις ε, συνεδριάσεις αυτών των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, διεθνών οργανισμών, για να μην κάνουμε δηλαδή την ίδια δουλειά δέκα φορές για την ανάλυση των σχεδίων διότι εμείς κάλλιστα μπορούμε να βασιστούμε είναι η mutually reliance δηλαδή να βασιζόμαστε στο σχέδιο το οποίο έχει κάνει μια, ένας άλλος οργανισμός αυτό μας μειώνει το κόστος διότι πολλές φορές εμείς συγχρηματοδοτούμε ένα σχέδιο και ο δανειζόμενος μάλλον και ο δανειστής θα έπρεπε να έχει μία, μία ενιαία ανάλυση με τους άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση και όχι μία ανάλυση για τον κάθε οργανισμό. Πέμπτο σημείο που αναφέρατε είναι το blending. Δηλαδή να συνδυάζουμε δάνεια και επιδοτήσεις. Για να έχει δηλαδή μεγαλύτερη πρόσβαση σε προτιμησιακά ταμεία ή ΕΤΕ. Το αναφέρατε εσείς, είναι το εγκυτικό ταμείο για τις υποδομές στην Αφρική, όπου συνδυάζουμε δάνεια της ΕΤΕ με επιδοτήσεις ε, που προέρχονται από αυτό το ταμείο που χρηματοδοτείται και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και από εκούσιες εισφορές των κρατών μελών. Και ε, συνδυάζουμε μαζί με αυτό το Εγγυητικό Ταμείο Λοιπόν, μαζί με άλλες ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, ναι, σύμφωνοι στο blending για τα δάνεια της ΕΤΕ σε συνδυασμό με άλλου είδους επιδοτήσεις και εισφορές. Άλλο που θέσατε κύριε εισηγητά είναι το θέμα των οροφών. οι τωρινές οροφές μας δημιουργούν πρόβλημα, διότι τα κράτη-μέλη όταν ξέσπασε η κρίση μας ζήτησαν να επιταχύνουμε τη χορήγηση δανείων όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός. Δηλαδή εμείς χρησιμοποίησαμε τους χρηματοπιστωτικούς μας φακέλους πολύ πιο γρήγορα. Οπότε το διαθέσιμο ποσό που έχουμε σήμερα είναι περιορισμένο, αν όχι μειωμένο. Πιο συγκεκριμένα στο κονδύλι για τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή τις χώρες που βρίσκονται στα πρόθυρα της προσχώρησης. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μία λύση, διότι εμείς αναγγείλαμε σε αυτές τις χώρες που είναι και πιο κοντινές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αναγγείλαμε ότι θα γίνετε μέλη και ξαφνικά στο απότομα σταματάμε όλες μας τις δράσεις σε αυτές τις χώρες πρέπει να βρούμε μια λύση. Αν λοιπόν επιπλέον μας ζητήσουν να παρέμβουμε και σε άλλες χώρες και αναφέρω εδώ πέντε χώρες που θα πρέπει, στις οποίες θα πρέπει να παρέμβουμε στο μέλλον ε, πρέπει να προσαρμόσουμε αναλογικά και την οροφή για τις ε, παρεμβάσεις μας σε αυτές τις χώρες. Επίσης τελευταίο σημείο κύριε Σιγητά αναφέρατε τις μελλοντικές δημοσιονομικές προπτικές που θα αρχίσουν το, 2014. Η συζήτηση πρέπει να αρχίσει σύντομα, διότι θα πρέπει να ξαναδούμε όλη τη διάρθρωση της ε, χρηματοπιστωτική, του συστήματος χρηματοπιστωτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπό το φως αυτών των χρηματοπιστωτικών των δημοσιονομικών συγγνώμη, προπτικών θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε ορισμένες από τις ε, ιδέες που ετέθησαν επί τάπητος. Αυτά κυρία Πρόεδρε για τις πρώτες ιδέες του συγκητή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μεγάλη σύμπτωση απόψεων. Ρωτώ τώρα την αίθουσα, θέλει κανείς το λόγο. Ο Γιώραν. Μία ερώτηση για να δω αν κατάλαβα καλά από τους δύο μιλητές μας. Αν τα κράτη-μέλη διστάζουν να παραταθεί η εντολή της ΕΤΕ. Είναι ουσιαστική φύση αυτή η αντίρρηση ή φοβόνται το κόστος διαβλέπουν κάποιο κίνδυνο. Αν επεκταθεί ή παραταθεί εξωτερική εντολή είναι πιο δύσκολο να δώσουν και μεγαλύτερο ρόλο της στην ΕΤΕ στο εσωτερικό της Ένωσης. Σχολιάστε το. Γιατί αυτή η αντίσταση. Είναι ουσιαστική ή πρακτική οικονομική η λογη Ευχαριστώ η Χέλγα Τρίπολα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση κύριε Μέιστατ και σας ε, θα ευχαριστήσω και τον κύριο Κάλ, Κάλφαν. Υποστηρίζουμε, θέλω να τονίσω, την γραμμή που ακολουθείτε. Θα ήθελα όμως τώρα να σας υποβάλω το εξή. Λέτε ότι η ανάγκη χρηματοδότησης της ε, ΕΤΕ με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των χωρών όπου λαμβάνει η χώρα η ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αναφέρεται στο εκτελεστικό κομμάτι και όχι μοναχά στο προήμιο της απόφασης. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας να το τονίσουμε αυτό. Επίσης και η αηφόρος διαχείρισης των παγκοσμίων πόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 της συνθήκης, θα πρέπει να αναφέρεται και στην απόφαση αυτή. <coughs> Γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει μεγαλύτερη επίπτωση και έμφαση στις μέρημνες για το περιβάλλον και την αηφορία. Θα ήθελα λοιπόν να τεθεί σε ένα πιο προεξάρχον σημείο στο κείμενο. Δεύτερον, η διατύπωση για την διαβούλευση ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί. Τρίτο σημείο. Η ΕΤΕ θα πρέπει να έχει σαφή κριτήρια αποκλεισμού επί τη βάση ε, κριτηρίων αηφορίας και περιβάλλοντος. Και στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται μια ανεξάρτητη αξιολόγηση σε επιπτώσει για το περιβάλλον προτού ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ. Θα σας δώσω και άλλα στοιχεία, άλλες ε, ε, προτάσεις από μια πράσινη οπτική γωνία. Σας υποστηρίζουμε λοιπόν πάρα πολύ, αλλά ο στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση ως μια σημεία, ώστε μπορούμε να καταλήξουμε και σε μια συμβαστική λύση. Α, ωραία, ο Καλ. Μερικά σύντομα σχόλια. Πρώτον, ευχαριστώ τον εισηγητή για την φιλόδοξη δουλειά του. Άριστη δουλειά. Πήγε σε βάθος στο θέμα αυτό. όταν μπαίνει κανεί σε βάθος στην ουσία υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει στο επίπεδο της μικροδιαχείρισης. Και πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία. Ας μην είπε ο φίλος μας από την ΕΤΕ είναι ευχαριστημένος, δεν έχω αντίρρηση. Συμφωνούμε με τη μέθοδο του εισηγητή, συζητήσαμε τα θέματα και την προηγούμενη εβδομάδα, υποβάλαμε και τροπολογίες, θα υποβάλουμε άλλες τροπολογίες το θέμα είναι πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ως εργαλείο να υποστηρίξει άλλες σημαντικές αποφάσεις της Ένωσης όπως στρατηγική του 2020, στρατηγική για τη Βαλτική, μακροστρατηγική, στρατηγική για το Δούναβι, Αυτά θα τα θέσουμε σε μορφή τροπολογιών. Είμαι σίγουρο ότι τελικά η έκθεση θα είναι πάρα, πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ η Βάρβαρα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σταθώ στην poverty reduction. Για να συμβεί κάτι τέτοιο όπως το, το ανέφερε και κάποιος ε, προλαλεί σας, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προσωπικού και πόρων. Ξέρετε ότι υπάρχει βέβαια κρίση σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν μπορεί λοιπόν να ονειρεύεται μακρόπνοα ή ετε, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία έμεση προσέγγιση να ασχολείται δηλαδή με σχέδια τα οποία έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στον πληθυσμό, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, ε, καταπολέμηση της φτώχειας και τα λοιπά και αυτό και μέσα στο εσωτερικό της Σούρε Κόμιτη. Ευχαριστώ. Κύριε Μέιστατ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το λόγο για την αντίσταση που βλέπουμε από ορισμένε χώρες στην ιδέα του να επεκταθούν οι δραστηριότητε τη ΕΤΕ εκτός της Ένωση, μετατρέποντα κατά κάποιο τρόπο την ΕΤΕ σε μια πραγματική τράπεζα ανάπτυξη είναι δυτή. Πρώτο είναι ο φόβος και το είπανε ανοιχτά μερικές χώρες αν αυξήσει τη δράση της εκτός της Ένωσης η ΕΤΕ αυτό είναι σε βάρος της δράσης της στο ιστορικό της Ένωσης και μερικές χώρες μέλη χρειάζονται την ΕΤΕ μέσα στην Ένωση ιδιαίτερα όσον αφορά τη στρατηγική του 2020 για σημαντικές στρατηγικές στην Ένωση όπως στρατηγική για τη Βαλτική και το Δούναβι. Ο φόβος λοιπόν είναι αν η ΕΤΕ επεκταθεί πολύ εκτός της Ένωσης αυτό να είναι σε βάρος της δράσης στο εσωτερικό. Ο δεύτερος λόγος αντιστάσεων είναι το ότι μερικές χώρες μέλη έχουν δική τους εθνική υπηρεσία αναπτυξιακού χαρακτήρα και δεν θέλουν ανταγωνισμό εντός εισαγωγικών εκ μέρους μιας ενός οργάνου της Ένωσης. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι γιατί το δεν υπάρχει τόσο ευρεία ομοφωνία για τη δράση εκτός της Ένωσης. Αντίθετα υπάρχει ευρεία συνένεση για δράση εντός της Ένωσης. Δεν παίρνω θέση για τις τροπολογίες, αλλά όντως ορισμένες ιδεολογικές σκέψεις να μπουν στο κείμενο της απόφασης μπορεί να ληφθεί υπόψη γιατί όχι. Η τελευταία ερώτηση προς την τελίδα Ευρωβουλευτή το να παίξει μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο η ΕΤΕ. Ναι, αν αυτό μας επιτρέπεται με τα εργαλεία που έχουμε που δουλεύουν με το επιτόκιο της αγοράς. Η εμπειρία μας μας δείχνει ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε δράσεις σημαντικής κοινωνικής, κοινωνικού χαρακτήρα σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης κλπ. Εξαιρέσεις υπάρχουν. Ε. Χρηματοδοτήσουμε ε, νοσοκομεία. Αλλά είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους προγράμματα με δάνεια που έχουν κόστος. Διότι η επιστροφή γίνεται με βάση επιτόκιο αγοράς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλου είδους εργαλεία και όχι δάνεια της ΕΤΕ. Äh, πέντε λεπτά ακόμα έχουμε. <laughs> Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για την τροπολογία 55. Ποιος είναι ο λόγος για να υπάρξει αυτή η αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο. Συνδέεται παράτημα 1 τροπολογία 55 έχει να κάνει κάτι με το παράρτημα 2 ή γενικά με τις δραστηριότητες η αύξηση αυτή. Και δεύτερον, ποιο είναι το επίπεδο των αποθεμάτων σε ποσοστό για τα, ε, για τα δάνεια τα οποία θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα. Ποια είναι τα, ποια είναι τα αποθέματα που έχετε για δάνεια χαμηλού επίπεδου, είναι μηδενικά, είναι χαμηλά, πόσα είναι. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Για το δεύτερο αυτό ερώτημα, ναι, πράγματι. Εφαρμόζουμε τους κανονικούς, τους συνήθεις κανόνες για μια τράπεζα, τις ε, απαιτήσει της Βασιλείας. Πρέπει επομένως ένα τμήμα του κεφαλαίου μας να χρησιμοποιείται ως αποθεματικό για να καλυφθούν επικίνδυνες δανειοδοτήσεις, οι οποίες απαιτούν περισσότερη κάλυψη σε κεφάλαιο. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο εμεί είμαστε σε συζήτηση με την Κομισιόν. Είχα μια συνάντηση με την Κομισιόν σήμερα το πρωί για τη στρατηγική 2020 τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και την ανάγκη να εξεύρουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα έδιναν μια καλύτερη μόχλευση στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά συγχρόνως θα μείωναν την ανάγκη να υπάρξει κατανάλωση κεφαλαίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ποσοστό που έχουμε για τα δάνεια αυτά που αναφέρατε είναι αυτή τη στιγμή 0,4% για τα δάνεια τα οποία είναι επικίνδυνου χαρακτήρα. Επομένως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις δανειοδοτήσεις της ΕΤΕ. Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, για να κλείσουμε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα απλώς εν συντομία να δώσω μερικές απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία ετέθηκαν. Έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και ξέρουμε ότι η δραστηριότητα της ΕΤΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 10% των συνολικών δραστηριοτήτων τους ότι επομένως αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει το ρόλο της τράπεζας μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να σταθεί σαν επιχείρημα όταν αναφερόμαστε στην ε, επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι το θέμα του προϋπολογισμού το οποίο ευαισθητοποιεί, για το οποίο είναι πολύ ευαίσθητες μερικές χώρες ε, μέλη το ερώτημα του κυρίου Γκουτμάνης. Ανέφερε ο κύριος Μέστατ ότι η συνολική έκθεση σε επικίνδυνα δάνεια της τράπεζας είναι πολύ χαμηλή. Αλλά εδώ είναι ειδική περίπτωση το έγγραφο που, που εξετάσουμε. Γιατί αυτές είναι οι δανειοδοτήσεις της τράπεζας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με εγγύησεις Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο δυνατότητες, είτε να αναλάβει μόνη της τον κίνδυνο, οπότε είναι πάρα πολύ ε, αυστηρές οι προϋποθέσεις για να διατηρήσει το υψηλό rating που έχει η τράπεζα, την υψηλή της βαθμολογία. Και δεύτερον, υπάρχουν δράσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να γίνουν ίδιο κίνδυνο της τράπεζας και καλύπτονται με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εγγύηση γίνεται από ένα ταμείο εγγύηση το οποίο το διαχειρίζεται η ίδια η τράπεζα και το οποίο καλύπτει το 9% της συνολικής εγγύησης που καλύπτει μέχρι 65% των ενεργειών της τράπεζας. Αν δείτε λοιπόν πόσα χρήματα έχει αυτό το ταμείο, μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ σημαντική μόχλευση για τις δραστηριότητες της τράπεζας της ΕΤΕΚΤΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ακόμα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, το οποίο έθεσε και η Helga Triple. Αυτό είναι οι επιτόπιες διαβολεύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και υπάρχουν πολλές απόψεις που έχουν διατυπωθεί. Ο πρώτος Μέισταν δεν το ανέφερε, αλλά η τράπεζα έχει αυτούς οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι οι υποστηρικτές των προγραμμάτων της, κράτη ή φορείς που επομίζονται την ε, διαχείριση ενός ε, Ενό σχεδίου. Υπάρχει αυτό λοιπόν ο οποίο προωθεί τη δανειοδότηση και αυτό το οποίο ζητούμε εμείς από την ΕΤΕ είναι να απαιτεί από αυτούς που επομίζονται τη διαχείριση του δανείου να αξασφαλίσουν ότι γίνονται και τοπικές διαβουλεύσεις. Δεν είναι η τράπεζα λοιπόν, αλλά είναι οι φορείς αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τη διαδικασία και υπάρχει βέβαια και το θέμα του να έχουμε μια πληρέστερη πληροφόρηση στο ίντερνετ ώστε να γνωρίσουν όλοι τι ακριβώς ε, γίνεται. Φυσικά αυτό μέσα στα όρια του ότι μπορεί να αποκαλυφθεί σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές αυτές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω πάλι σε όλους. Εάν δεν το έχετε κανονίσει ήδη, οι τροπολογίες μέχρι τις 29 Οκτωβρίου ώρα Παρασκευή και ημέρα 12 η ώρα το μεσημέρι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο σημείο. Κύριε Μέιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και σίγουρα θα ξαναβρεθούμε όταν συζητήσουμε για το θέμα της ατζέντα 2020. Μα ήρθε ο Ράιμερ Μπέγγε, ο εισηγητής μας ο οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Πρέπει να τα κάνουμε λοιπόν και τα δύο. Πρέπει αμέσως να περάσουμε στον διορθωτικό προϋπολογισμό. Είναι το σημείο 5, αλλά και το σημείο 7 που έχει να κάνει με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε ίσως να συζητήσουμε τα δύο αυτά σημεία μαζί. Θα πρέπει να ξελαχανιάσει καταρχήν ο Ράιμερ και να καθίσει να ανοίξει το μικροφωνό του και να μας κάνει μία εισαγωγή στα θέματα αυτά. Θες να κάνεις ε, πρώτα μια εισαγωγή Λάσλο ή να ακούσουμε το Ράιμερ, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίσει και τα δύο θέματα. Είσαστε ουσιαστικά, ε, μπορείς, να μας πεις εσύ τι θέλεις μετά και να μιλήσεις προηγουμένως στο Ράιμερ. Εντάξει, συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που έχω καθυστερήσει λιγάκι. Έβαλνε χώρο στο Βερολίνο μία συζήτηση για τα θέματα τα, τα δημοσιονομικά που περιλαμβάνει ακόμα και τη συζήτηση των ιδιών πόρων. Και φαίνεται ότι βράζουν τα πράγματα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά την ε, διαθεσμική συμφωνία, τη βάση διαθεσμικής συμφωνίας 7 ε, Μαΐου 2006 πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το πολύ ένα δισεκατομμύριο μπορούν να κινητοποιηθούν ετησίως. Η Κομισιόν μετά από την αίτηση της Ιλλανδίας λόγω των περιφερειακών αυτών πλημμυρών του 2009 και επί τη βάση των στοιχείων που έχει δοθεί, έχουν δοθεί από την Ιρλανδική πλευρά για το ύψος των ζημιών ζήτησε την εφαρμογή του, της ειδική ρήτρας του άρθρου 2.2 βάσει της οποίας μπορούν να συμπεριληφθούν και περιφερειακού χαρακτήρα καταστροφές στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης και να μπορεί να επέμβει το Ταμείο Αλληλεγγύης. Εδώ λόγω της σοβαρότητας αυτής της περιφερειακής καταστροφής μπορεί βάσει του κανονισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης να παρέμβει το Ταμείο και αυτό ζητάει η Κομισιόν να υπάρξει λοιπόν παροχή βοήθειας βάσει αυτής της ρήτρα. Πρόκειται για 13 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης που προτείνεται να δοθούν. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, εξάλλου αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Σας πεθυμίζω ότι πριν από την ψηφοφορία θα πρέπει να ακούσουμε και την άποψη της Περιφερειακής Επιτροπής και βέβαια έχουμε το πρόβλημα ότι οι πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να προέλθουν από το κοινωνικό ταμείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται μονίμως στην μέση διάταξη σε σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης και την ανάγκη να χρησιμοποιήσει πόρους από το κοινωνικό ταμείο εάν δεν έχει το ίδιο απαραίτητους πόρους. Αυτό είναι το μόνο σημείο το οποίο πρέπει να σας ε, αναφέρω και κατά τα άλλα υποστηρίζω αυτή την πρόταση στο όνομα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα νέα της Κομπού αναφέρεται ότι η προθεσμία τροπολογιών είναι το μεσημέρι της 28 Οκτωβρίου 9 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε και στη δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου θα έρθει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Αλλά αν δεν μας δώσει ο Λάζο τα χρήματα δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε. Δεν χρειάζεται να φοβάστε λέει ο Λάσλο γιατί είναι απόλυτα σαφές ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η Επιτροπή Προϋπολογισμών πάντα υποστηρίζει τη χορήγηση αυτής της βοήθειας και ο εισηγητής σας το υποστηρίζει εδώ, ακόμα και αν είναι ζημίες περιορισμένες σε περιφερειακό μονάχα επίπεδο. Στη χώρα μου υπάρχουν πολλοί ευρωσκεπτικιστέ οι οποίοι συζήτησαν για το θέμα αυτό, γιατί και εμείς στην Ουγγαρία είχαμε μια μεγάλη καταστροφή με την δηλητηριώδη ε, λάσπη, την κόκκινη λάσπη, η οποία είχε περιορισμένο γεωγραφικό χαρακτήρα, αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Εμείς βρισκόμαστε πάνω από το 0,6% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά εφόσον έχουμε μια... Αυτό που είναι κάτω από το όριο βέβαια είναι η φυσική καταστροφή Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση, επειδή έχουμε μια φυσική καταστροφή και όχι μια βιομηχανική καταστροφή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο λείπει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, αυτό θέλω να τονίσω και για την τροπολογία υπαριθμών 9 εγώ την υποστηρίζω ως εισηγητής, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Ότι υπάρχουν και άλλες δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν από βιομηχανική ρήπανση, παραδείγματος χάρη όπως αυτή της Ουγγαρίας, οι οποίες μπορεί να είναι ε, πάρα πολύ σοβαρές, παραδείγματος χάρη καταστροφές όπως αυτές που είχαν λάβει στο παρελθόν στην Ινδία, δηλητήριαση μεγάλου μέρους του πληθυσμού η βασική αρχή είναι ότι αυτός ο οποίος δημιουργεί τη ρήπανση θα πρέπει και να πληρώνει. Ίσως λοιπόν στο μέλλον θα πρέπει να είναι λογικό να έχουμε μια ειδική υπηρεσία η οποία να δίδει δανειοδότηση για άμεση δράση, όχι μονάχα μερικούς ε, μήνες αργότερα, ώστε να βοηθηθούν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά η, όταν καταλογιστεί η ευθύνη, θα πρέπει ο υπεύθυνο να πληρώσει το κόστος. Ωραία, λοιπόν, οπότε έχει κλείσει το θέμα αυτό. Η καταληκτική προθεσμία είναι πάλι 28 Οκτωβρίου. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρχουν τροπολογίες. Και η τελευταία μου παρατήρηση που είναι κάπως παράλληλη. Εγώ σοκαρίστηκα στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα όταν η συγγήτριά μας η Συντόνια είχε τέσσερα λεπτά για να λάβει το λόγο για όλο τον προϋπολογισμό και εγώ απλώς μπόρεσα να αναφερθώ σε ένα μικρό θέμα τον διορθωτικό προϋπολογισμό είχα και εγώ τέσσερα λεπτά. Κάτι δεν πάει καλά στην οργάνωση του χρόνου ομιλίας μας. Και πραγματικά έριξα το φταίξιμο και στον εαυτό μου. Γιατί για ένα τόσο σημαντικό θέμα να έχει τέσσερα λεπτά η συγγήτρια η οποία εργάζεται για ένα χρόνο για το θέμα αυτό και για ένα κούτσικο θέμα όπως ήταν το δικό μου να δίνουμε τέσσερα λεπτά όταν δεν χρειάζεται καν ο εισηγητής αυτού του θέματος να λάβει το λόγο. Και ήταν παράξενο αυτό γιατί είχα δύο διορθωτικούς προϋπολογισμούς Τέσσερα λεπτά, συν τέσσερα λεπτά, συν χρόνο στη συνέχεια για να κλείσω τη συζήτηση. Νομίζω θα πρέπει να θέσουμε αυτό το ζήτημα και να τονίσουμε ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τα βασικότερα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να δίνουμε στον εισηγητή ή στην εισηγήτρια να δίνει στην ε, δημοσιότητα την ουσία του προπολογισμού και όχι να δίνουμε τέσσερα λεπτά για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Πέντε λεπτά μίλησα τώρα, αλλά στην Ολομέλεια δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τόσο χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Λάσλο. Όλα αυτά λοιπόν τα κατανοούμε, αλλά η διοίκηση του Κοινοβουλίου χρησιμοποίησε την πάγια διαδικασία ο εισηγητής έχει τέσσερα λεπτά, ανεξάρτητα από την ε, σημαντικότητα του θέματος το οποίο πρέπει να διεξέλθει ή αν. Να υποστηρίξω κι εγώ μερικές από τις παρατηρήσεις του Λάσλο. Όντως χρειάζεται χρόνος για να φτάσουν τα χρήματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μερικοί από εμάς δυσπιστούμε για την ιδέα αυτή του Ταμείου Αγγελεγγύης. Όταν είχαμε τις πλημμύρες στις Άλπες, θυμάμαι τους ε, Γερμανούς που είπαν μην το κάνετε γιατί θα πληρώνετε για τα επόμενα 25 χρόνια και μάλλον αυτό συμβαίνει. θέτω το ερώτημα αυτό, μιας και έχουμε εκπροσώπους της Κομισιόν. Για το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί τα πράγματα να κινηθούν πιο γρήγορα στο μέλλον ή οι κανόνες ορίζουν ότι χρειάζεται τόσο πολύς χρόνος. Και δεύτερο, κάτι που είπε ο Λάσλο όχι θεομηνίες αλλά άλλου είδους καταστροφές που συζητήθηκαν όταν συζητούσαμε για το Ταμείο Εκλεγγύης Τι δυνατότητα υπάρχει όμως χάρη για την καταστροφή στην Ουγγαρία και το Ταμείο Εκλεγγύης Τι μπορεί να γίνει Κρόλη Ευχαριστώ Ευχαριστώ τον συγκητή και τον ενθουσιασμό σχετικά με τα κονδύλια του Ταμείου Ελληνικής. Η πόλη από την οποία προέρχομαι είχε πλημμύρα το 2009 18 εκατομμύρια στελγίνες είχα μόνο στο σπίτι μου. Σε ιδιωτικές οικίε, μάλλον. Και πολλές ε, βιομηχανίες στην πόλη πλήγησαν επίση. Ήταν σημαντικό το ότι δόθηκαν τα λεφτά, γι' αυτό έχω συγκεκριμένο συμφέρον, αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξή. Όχι αμέσως. Όπω είπε ο Λάσλο, σωστά, θα πρέπει να δούμε μήπω τυχόν κάποιο άλλο είναι υπεύθυνο. Άρα να φέρει και ένα τμήμα της ευθύνη. Αν το επιταχύνουμε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Βέβαια, αυτό που είπε ο Λάσλο για ένα μηχανισμό δανείου για ε, καταστροφές που προέρχονται από χέρι ανθρώπου υπάρχει άμεση ανάγκη καθαρισμό, άρση του προβλήματος για την υγεία των κατοίκων αυτό ξεπερνάει την, της συνήθη δράση των υπηρεσιών. Αυτό θα έπρεπε να προβλέπετε κάπου. Επαναλαμβάνω, συμφωνώ με τον Λάσλο. Είναι γελίο αυτός που παρουσιάζει την έκθεση για τους προπολογισμού για το κοινοβούλιο, να δίνει 135 δις και να του δίνει μόνο 4 λεπτά ομιλίας, ξέρω από εμπειρία, αν στη διάσκεψη των Προέδρων, αν το φέρεις αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων, μία ώρα θα δινόταν στον εισηγητή και για στους άλλους εισηγητούς επιπλέον. Πρόεδρος, ο για να κλείνουμε. Ευχαριστώ τον Λάσλο και όλους για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουν ξεκινήσει. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης υπάρχει και το άρθρο 120 το οποίο έχει τύχει κακομεταχείρισης βέβαια αλλά το οποίο όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα λέει ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει μία βοήθεια. Βάσει αυτού του άρθρου το Κοινοβούλιο μπορεί να πληροφορηθεί για τη χρήση αυτού του μηχανισμού. Επίσης, η Κομισιόν έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν το άρθρο 122 για την χρήση σταθεροποιητικών μηχανισμών για να αντιμετωπιστούν καταστροφές σε τραπεζικό ή και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Λοιπόν, η Κομισιόν δεν έχει πρόβλημα να είναι καινοτόμα σε τέτοια ζητήματα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Σούριαν, μονάχα μια φράση η Σιδονία δεν μου είπε τίποτα για, τα, <laughs> για το χρόνο που καταδαπάνησα. Ε, εντάξει, έτσι φανταστήκαμε και εμείς ότι θα έκανε. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία, την 5η στις 12, όπως είπαμε προηγουμένως, ξανά έχουμε πρόεδρο και του ξαναδίνω την διαχείριση της συνεδρίασης. Ευχαριστώ Γιούτα. Συγγνώμη, θα ζητήσω και συγγνώμη στον πρόεδρο Μέιστα, διότι ε, ήμουν υποχρεωμένος να προεδρεύσω έναν, σε έναν τρίλογο για τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Και αυτό δεν θα στοιχήσει ούτε ένα ευρώ λοιπόν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης ο Τζοβάνι Λαβία, ο εισηγητής, είναι εδώ. Αναβάλλεται το σημείο. Ο Τζοβάνι δεν είναι εδώ, μας είχε πει λοιπόν ότι αναβάλλεται, εξαφανίστηκε λοιπόν με το σημείο του ο Τζοβάνι. Ο κύριος Αλφόνση μας ζήτησε ότι θέλει μια διαφορετική διαδικασία. αγαπητέ Μα τι έχει αυτό το μικρόφωνο, τίποτα, τίποτα δεν είχε εντάξει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να αποφασίσουμε για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την αλληλευτική πολιτική και τον τομέα του δικαίου της θαλάσσης. Λοιπόν, δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτή η πρόταση, είναι τεχνικά τα θέματα, η Επιτροπή λοιπόν δεν έχει αντιρρήσεις εγώ θα έλεγα δε η Επιτροπή Ελίας ε, η οποία ήταν και αρμόδια επί της ουσίας, εκφράστηκε για τις μετροπολογίες, δεν είχε καμία αντίρρηση. Προτείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε να πληροφορήσετε την αρμόδια επιτροπή λέγοντας ότι επειδή δεν υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις ε, περνάει αυτή η πρόταση και επιτρέπει και τις διατάξεις να ισχύσουν γρηγορότερα. Λοιπόν, έχετε τίποτα να πείτε, σχόλια, παρατηρήσεις, αν όχι. Ακολουθούμε τη σύσταση του εισηγητή. Και θα στείλουμε μια επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Στη συνέχεια πάμε στο επόμενο σημείο. το σημείο 10. Το 10. 11, 12, 13, 14, 15. Κοινή συζήτηση για πολλά σχέδια κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Και η Μπάρμπαρα Ματέρα είναι η συγγήτριά μας. Λοιπόν, Μπάρμπαρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακαλώ τους συναδέλφους να με ακούσουν διότι ήρθαν στην Επιτροπή μας έξι αιτήματα για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και έρχονται όλες από την Ολλανδία. Πρόκειται λοιπόν για τομείς που έχουν πληγεί από την κρίση, είναι ο υφαντουργικός και αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας. Η το πρώτο μέτρο αφορά στην απόλυση 58 εργαζομένων της περιοχής Nord Holland και Ζουίτ Όλαντ, δηλαδή Βόρεια και Νότια Ολλανδία. Ζήτω συγγνώμη για την προφορά μου. Πρόκειται για 2.220.000 ευρώ πάνω κάτω. Πάντοτε λοιπόν στο γραφικό τομέα έχουμε εδώ 720 σε 79 που ανήκουν σε 79 επιχειρήσεις στον τομέα της αναπαραγωγής μουλτιμέδια υλικού στην Νόρντ Όλαν και Ούτρεκτ, Βόρεια Ολλανδία και Ουτρέχτη. 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Μετά έχουμε 121 εργαζόμενους, 70 επιχειρήσεις, ποσό 2.890.000 ευρώ πάνω κάτω. Τέταρτο αίτημα. για 750 εργαζόμενους σε 45 επιχειρήσεις στο Τζέντερλαντ και αυτό πώς να το προφέρω αλήθεια πώς να το προφέρω δεν ξέρω αν προφέρεται Χόβερ Ίσελ λοιπόν για 2 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία, τα δύο τελευταία αιτήματα τα έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2 στο γάμα του κανονισμού όπου γίνονται δεκτές οι αιτήσει για την υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων. Και δίνονται λοιπόν αυτά τα κονδύλια και τα δέχθηκε η Επιτροπή διότι θεωρείται ότι αυτές οι απολύσεις θα επιβορυβαρύνουν στον κοινωνικό ιστό. Υποστηρίζονται λοιπόν 129 εργαζόμενοι που απολύθηκαν από 9 επιχειρήσει από το Λίμποργκ, το Λιμβούργο δηλαδή, με 550, α λάθος λάθος, 550.000 ευρώ, συγγνώμη, το τελευταίο λοιπόν αίτημα αφορά σε 140 εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε δύο επιχειρήσεις της περιοχής του Ντρέμπτεν με 450.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά τις προτάσεις που έγιναν Έψαξε να βρει budget line, λέει ο μιλήτρια, από ποσά τα οποία είχαν μείνει στο αποθομητικό. Πάντοτε ξέρω ότι οι, συναδέλ, συνάδελφοι περιμένουν από μένα να βρίσκω περιθώρια και όπου μπορεί να τραγανίσει η Κομισιόν, έτσι το λέω εγώ, Ρωσικιάρε. Ε, και ευελπίζουμε ότι στην 1η του Νοεμβρίου θα μπορέσουν να περάσουν αυτές οι εκθέσεις. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή την αίθουσα δύσκολα μπορώ να περασουν αυτέ οι εκθέσει. ευχαριστω αγαπητοι συναδελφοι ειναι εδω η ευρωπαικη επιτροπη σε αυτη την αιθουσα δυσκολα μπορω να εντοπισω Α, ο Γενικό Διευθυντή είναι εδώ. Μα πραγματικά ε, τα έχω εντελώ ε, χαμένα. σα έχουν βάλει στο βάθο τη αίθουσα σαν του κακού μαθητέ στο Δημοτικό. Αλλά επειδή εδώ είμαστε στην αίθουσα συνδιαλλαγή, είστε μεταξύ των καλών μαθητών. Λοιπόν, ο αρμόδιος από τη Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτά που είπε η εισηγήτριά μας. Θέλετε να συμπληρώσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια μονάχα παρατήρηση. Οι υποθέσεις αυτές είναι όπως, όπως είδατε περίπου ταυτόσιμες γιατί αφορούν τον ίδιο τομέα και το ίδιο βασικό πρόβλημα απολύσεων. Για λόγους όμως που πηγάζουν κατευθείαν από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, εμείς πρέπει να τις παρουσιάσουμε βάσει του άρθρου 2β σαν περιφερειακές περιπτώσεις ή σαν έκτακτες περιπτώσεις βάσει του άρθρου 2C. Γι' αυτό έχετε έξι περιπτώσεις και όχι μια μεγάλη, μεγάλη περίπτωση. Κατά τα άλλα νομίζω ότι η συγγήτρια έχει δώσει μια πλήρη εξήγηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρέμπια λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται λοιπόν για ένα αρκετά σημαντικό πακέτο. Έχουμε έξι διαφορετικές περιπτώσεις από οι οποίες βγαίνουν από δύο διαφορετικές διαδικασίες, τέσσερα συν δύο. Είναι τρεις χιλιάδες εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί Αν δεν υπάρχουν λοιπόν άλλοι ετούντες το λόγο, θυμίζω λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα η Επιτροπή Απασχόλησης θα γνωμοδοτήσει. Προθεσμία για τις 8 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι, μεθαύριο δηλαδή, και θα εγκρίνουμε τις εκθέσεις της κυρίας Ματέρα στις 9 Νοεμβρίου για να περάσουν φυσικά από την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, πάμε στο σημείο 16. Το σημείο 16 είναι ένα σημείο πάρα πολύ τεχνικό υπερβολικά βαρετό σύμφωνα με την διαθεσμική συμφωνία πρόκειται για διορθώσεις που είναι υπό την αρμοδιότητα της Κομισιόν και η αρχή του προϋπολογισμού απλώς ε, ενημερώνεται. Τώρα, αν ο Ράιμερ Μπούγκε θέλει να, απλώς να κάνει μια ανακοίνωση Όσο προειδοποίηση στην Κομισιόν δεν χρειάζεται καν να κάνουμε μια ξεσυρά ημερ. Τι Νομίζω ότι μπορούμε <clears throat> να καταγράψουμε αυτή την τεχνική προσαρμογή. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τεχνικών προσαρμογών που είναι απαραίτητες στην τεχνική του προϋπολογισμού. δεν είναι το είδος αλλαγής η οποία την χάνει διαπραγμάτευσης και διαμαχών. Είναι μια τεχνική προσαρμογή σε σχέση με τις ε, τιμές και το εθνικό εισόδημα που σημαίνουν και κάποιες τροποποιήσεις στην κατηγορία 1β βάσει της οποίας ε, υπολογίζεται στην κατηγορία 1β που πρέπει να υπολογίζεται <coughs> το συνολικό, το σωρευτικό ΑΕΠ από το 2007-2009. Εάν έχει αποκλίνει κατά πάνω από 5% από το ποσό που αναφερόταν στην ε, συμφωνία θα πρέπει να γίνει απαραίτητη αυτή η προσαρμογή. Είναι τρία κράτη-μέλη που αφορά αυτή η προσαρμογή, Πολωνία, Τσεχία και Σλοβακία και οι χώρες αυτές έχουν περίπου ένα, εκατομμύριο... ένα ένα δισεκατομμύριο σε υποχρεώσει και 228 εκατομμύρια σε πληρωμών για τα χρόνια 2011-2013. Αυτό λοιπόν είναι απα... απόρρια αυτής της ε, προσαρμογής και αυτό δείχνει και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι τεχνικέ προσαρμογέ και πρέπει πράγματι να λάβουμε γνώση αυτή τη αλλαγή και να περιοριστούμε εκεί. Τρέμπιεν λέω. Τροποποιώ λοιπόν, την πρόταση σε Παρότι το θέμα είναι ανιαρό, παίρνει ένα χαρακτήρα πάθος όταν μας το εξηγεί ο Ράιμερ. Ελπίζω ότι η Κομισιόν να μην θέλει να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες. Κανένα να ζητάει το λόγο. Όλοι βρισκόμαστε σε έκσταση. Και περνάμε στο επόμενο σημείο. Όχι το 17. Προτείνω να περιμένουμε λίγο να έρθει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας που υποπτεύει το πρόγραμμα ITER ενώ το 17 γιατί η παρουσία του θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συζήτηση για το ITER. Και αυτή τη στιγμή μιλάει για αυτό το θέμα στην Επιτροπή ΙΤΡΕ Άρα σε μερικά λεπτά θα μας έρθει και εδώ να τον περιμένουμε για το 17. Ας περάσουμε στο 18. Ξαναδίνω το λόγο στην Μπάρμπρα Ματέρα για ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Για την έκθεσή της σχετικά με την Ιρλανδία. Θέλει να μιλήσει. Όχι, όχι, απλώς ήμουν αφηρημένη για ένα λεπτό. Ήδη εμείς συζητήσαμε για την κινητοποίηση του Ταμείου για αυτό το αίτημα. Θέλοντας δηλαδή μπορούμε και να ψηφίσουμε. Αλλά επειδή λείπουν πολλοί συνάδελφοι, μήπως θα έπρεπε να ψηφίσουμε, να, αναβάλουμε την ψηφοφορία, εσείς πρόεδρε μου να αποφασίσετε. Έχουμε τη γνωμοδότηση της ψηφής Απασχόλησης, δεν έχουμε τροπολογίες, μπορούμε να ψηφίσουμε. Αν θέλετε να μας θυμίσετε κάτι, ναι, αλλιώς ψηφίζουμε. Ωραία, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Μπόρκος. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση. Μείον ο κακός κύριος Μπόκρος. Το γράφουμε αυτό για τα πρακτικά. Συνεχίζει η ψηφοφορία 19. Λάσλο Σουριάν θα μας προτείνει μια μεταφορά. Λάσλο. Δεν προτείνω εγώ τη μεταφορά, η Κομισιόν την προτείνει. Μια γενική μεταφορά. και θα πρέπει να είμαστε, να περήφανοι γιατί πριν από ένα χρόνο είπαμε ότι το ποσά για τον τίτλο 1β δεν επαρκούν. Να η πρόταση να αυξαθεί το 1β με παραπάνω από 1,1 δις ευρώ. Σημαντικό αυτό. Τα δέκα τελευταία χρόνια αυτή η πρόταση της Euro σε ευρώ είναι η πιο μεγάλη μεταφορά. Όχι σε ποσοστό. Πριν από πέντε χρόνια σε ποσοστό ήταν λίγο πιο μεγάλη. Σε ευρώ όμως όχι. Βέβαια δεν με παραικανοποιεί αυτή η πρόταση και θα σας εξηγήσω γιατί. Περικόπτουμε κονδύλια και αυξάνουμε κονδύλια. Και τελικά οι γραμμές όπου περικόπτουμε τώρα είναι μια δαπάνη που μας δίνει την εντύπωση ότι είναι το 100%. έτσι ώστε να μην μείνουν τα δαπάνη τα χρήματα στη γραμμή. Οπότε πρέπει να αναλύσουμε ποια γραμμή δαπανήθηκε σωστά στην εφαρμογή ενώ στην εκτέλεση. Δεν είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα τελικά νούμερα. Θα πρέπει να δούμε τι ψηφίσαμε στον προπολογισμό, τι εκτελέστηκε και μετά να κρίνουμε αν αυτή η γραμμή ή η άλλη γραμμή εκτελέστηκε σωστά με σωστά αποτελέσματα ή όχι. Τα τελικά λοιπόν ποσοστά ή το 100% δεν είναι πάντα σωστό. Βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος και γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν. Δεν είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες των γραμμών για τις οποίες δίνουμε τώρα από άλλες πηγές. Τι θα συμβεί στο Συμβούλιο αν γίνει η πρόταση, να βάλουν νέο χρήμα στις γραμμές αυτές. Παρά το ότι, όσον αφορά το 1β, έχουμε την δήλωση ότι αν οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες από τον προπολογισμό που ψηφίστηκε, οι χώρες μέλη είναι διατεθειμένες να πληρώσουν. Τώρα βλέπουμε ότι αποδίδει η γραμμή για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο πλεόνασμα η γραμμή για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Καλό πράγμα η ανάλυση, καλό πράγμα και η ψηφοφορία και ο συγγητής σας προτείνει να ψηφίσουμε αυτές τις ε, μεταφορές, να ψηφίσουμε υπέρ. Υπάρχει καιρό του ζήν, καιρό του θνίσκιν. Υπάρχει καιρό του ψηφίζει, καιρό του μη ψηφίζει. Έτσι έλεγε ο Έριχ Μαρία Ρέμαρ, αλλά τα είχε κλέψει από τη βίβλο. Ο κύριο Γκότμαν, πρέπει να κάνει κάποια σχόλια εδώ. Παρακαλώ. Πολύ, σύντο... σύντομα σχόλια, γιατί συζήτησε ήδη με τον κύριο Σουριάν. Είναι δυνατόν να ρωτήσουμε την Κομισιόν Άδε με το φάκελο 22, βλέπουμε απορροφητικότητα μηνιαία για τρία διαφορετικά ταμεία. Θετικό. Για το 1β στην αύξηση των χρημάτων για την Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Εκτέλεση προγραμμάτων έχει πετύχει την άριστη ταχύτητα το ερώτημα είναι γιατί το κοινωνικό ταμείο δεν έχει πετύχει την άριστη ταχύτητα κίνησης, γιατί αν δούμε τους πίνακες, απορροφητικότητα στην αρχή της πενταετίας μόνο 19%. Γιατί τα δύο ταμεία είναι καλά και το κοινωνικό ταμείο δεν είναι. Μόνη μου ερώτηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. έχουμε τη μεταφορά του αιώνα. Διότι από την αρχή του 21ου αιώνα τόσο μεγάλη μεταφορά συνολική δεν είχαμε. 1.792 εκατομμύρια. Και ο συγκητής μας χρειάζεται χρόνο για να διαμορφώσει γνώμη για τη μεταφορά αυτή. ο κ. Γκοτμάνης έχει και μια συμπληρωματική ερώτηση. μπορούμε να ορίσουμε στόχο να υποβάλουμε τη μεταφορά αυτή σε ψηφοφορία στις 9 Νοεμβρίου γιατί η προθεσμία είναι 11 Νοεμβρίου. Και μέχρι τότε η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις του εισηγητή και του συναδέλφου. Προτείνω λοιπόν να ε, περάσουμε στην τελική ψηφοφορία το σημείο 20 πριν έρθουμε στο ΙΤΑΡ. Ο, ο Γενικός Διευθυντής ήρθε. Το λόγο στον κύριο Βλαντιμίρ Μάνκα για δύο μεταφορές νομίζω. Βλαντιμίρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι συντομότατος. Δύο μεταφορές. Η μία, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, λόγω των αλλαγών σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τη μετατροπή δύο προσωρινών θέσεων σε μία προσωρινή και μία μόνιμη. Η άλλη πρόταση είναι να μειωθούν οι θέσεις 1 ανάλογα με βαθμούς. Τα δύο ουσιαστικά μεταφράνουν ουδέτερη όσον αφορά τον προπολογισμό. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον χρήματα. Και μάλιστα γίνεται εξοικονόμηση 270 ευρώ. Προτείνω να γίνουν δεκτές. Πρόεδρος. Παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Ψηφίζουμε υπέρ. κατά αποχές εγκρίθηκε ομόφωνα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Σε 9 του Κοινοβουλίου. Εδώ έχουμε το Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι έχουμε τη σύνταξη για ορφανά για την τα μέλη όταν πεθάνει ένας βουλευτής ή πρώην ευρωβουλευτής μπορούμε να το σχεδιάσουμε αυτό να το υπολογίσουμε και έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες εδώ από ό,τι είχε προβλεφθεί θα, θα χρειαστούμε 150.000 ευρώ για να καλυφθεί αυτή η γραμμή προτείνω να το δεχτούμε Πρόεδρος Ψηφίζουμε για τις χείρες μου ουσιαστικά εδώ. Mixed feelings, με ανάμεικτα συναισθήματα. Ποιο είναι υπέρ τη ψήφου αυτή που ο εισηγητή θα προτείνει να υπερψηφίσουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, ομόφωνα για τους χείρους και τις χείρε και για τον εισηγητή μας. Κύριε εισηγητά, άλλες μεταφορές όχι. Ωραία, τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Και γυρίζουμε στο 17. Πρόκειται τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που χρειάζεται το πρόγραμμα, το έργο ITER. Η Επιτροπή Προπολογισμών ήδη το συζήτησε το θέμα πολλές φορές και θα είναι ένα από τα στοιχεία διαπραγμάτευσης που ξεκινάει αύριο με το Συμβούλιο για τον προπολογισμό του 11 και τον διορθωτικό του 10. για τον οποίο ακόμα τα τρία όργανα δεν συμφώνησαν. Πριν ξεκινήσουμε όμως αυτές τις διαπραγματεύσεις, κρίναμε σκόπιμο να ακούσουμε την άποψη αυτού που είναι υπεύθυνο τη υπηρεσία τη Κομισιόν, Γενικό Διευθυντή, ο κύριο Σμιτ. Ο Ράμερ Μπέγκε, ο συγγητή μα, μήπω να κάνει μια εισαγωγή. Νομίζω δεν χρειάζεται. Και στην ε, τελευταία συνεδρίασή μας είχα αναφέρει τις παρατηρήσεις μου παρουσία του Γενικού Διευθυντή για τα θέματα αυτά και έθεσα το ερώτημα του αν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο η χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ που βασίζεται σε ένα διεθνές consortium εκτός από μία πολιτική ομάδα οι άλλες πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν καταρχήν το να βρούμε αυτήν τη χρηματοδότηση αλλά φυσικά αυτό δεν θα είναι τόσο απλό γιατί πρέπει να υπάρξει μια πρόταση ώστε να θέσουμε σε διάθεση 400 εκατομμύρια από την γραμμή του προϋπολογισμού της Γεωργίας και θα χρειαστεί και στη συνέχεια να κάνουμε μεταφορές πιστώσεων και από άλλους τομείς της ε, έρευνας για να καλύψουμε την απαραίτητη διαχείριση, την, την ε, χρηματοδότηση μάλλον και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του εγχειρήματο του ΙΤΕΡ. Φυσικά όλα αυτά ξεπερνούν το πλαίσιο του δημοσιονομικού το οποίο είχε καταρχήν προβλεφθεί για το σχέδιο ΙΤΕΡ. Πρέπει επομένω να αντιμετωπίσουμε και τις δομές διαχείρισης, την παροχή συμβουλιών από εμπειρογνώμονες στο ίτερ, να εξασφαλίσουμε ότι έχει μια καλύτερη λειτουργία το ίτερ. Γι' αυτό θέτουμε αυτά τα θέματα στην Κομισιόν. Και θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι και η διαδικασία η οποία λαμβάνει η χώρα στο, στους κόλπους του Συμβουλίου. Μιλάμε για μια χρηματοδότηση, πρόσθετη χρηματοδότηση 1,4 δισεκατομμυρίων. Παραμένουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίσουμε και από την πλευρά του ε, Συμβουλίου προτού εγκρίνουμε κάτι το οποίο προφανώς είναι απαραίτητο σαν αρχή του προϋπολογισμού να μπορούμε να το αιτιολογήσουμε και ενώπιον της κοινή γνώμης. Φαντάζομαι ότι τα ερωτήματα αυτά θα τα απαντήσει ο κύριος Σμιτ και στη συνέχεια με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Ωραία κύριε Ισηγήτα. Ο Σαλβαδό Γκαρίγα ζήτησε το λόγο. Εγώ προτείνω αυτοί που έχουν να θέσουν ερωτήματα στην Κομισιόν να το πράξουμε τώρα, ώστε να μπορέσει συνολικά να απαντήσει ο κύριος Γενικός Διευθυντής, ο James Ellis, ο Paul Rubik και ο Σαλβαδό. Σαλβαδό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ανήκω σε μια πολιτική ομάδα η οποία υποστηρίζει τα μάλα το σχέδιο ΙΤΕΡ. Εμείς συμφωνούμε πάρα πολύ με το γεγονός ότι το ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σχέδιο για το μέλλον της έρευνας στην Ευρώπη για να εξασφαλίσει τη βιομηχανική και επιστημονική μας ανταγωνιστικότητα στο μέλλον. Αυτό, όπως είπε ο συνάδελφος Πέγγερ, το οποίο είναι υποσυζήτηση, είναι ένα σύνολο από αβεβαιότητες οι οποίες παραμένουν ακόμα μέσα στο σχέδιο αυτό και επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε το γεγονός ότι και πάλι μια ελληματική πρόβλεψη χρηματοοικονομική πρέπει να την ε, πληρώσει η γεωργία. Δηλαδή την ύφη πρέπει να την πληρώσει την ύφη της λανθασμένης σχεδίαση ενός βιομηχανικού σχεδίου θα πρέπει να την πληρώσει η γεωργία. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο στο μέλλον. <clears throat> Μας λέει η Κομισιόν ότι είναι το τελευταίο έτος στο οποίο θα υπάρξει πλεόνασμα στη Γεωργία το 2010 που θα επιτρέψει να κάνουμε τέτοιου είδους ε, ενέργειες. Γιατί το 2011-2012 οι προβλέψεις για τον αγροτικό τομέα δεν μας επιτρέπουν να θεωρούμε δεδομένο ένα τέτοιο πλεόνασμα. Συζητήσαμε και είχαμε πει την τελευταία φορά ότι θα έπρεπε να ήταν η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιήσουμε τη γεωργία ως κορβανά από τον οποίο θα αντλήσουμε χρήματα και ότι δεν πρέπει στο μέλλον να χρηματοδοτούμε τέτοιες ενέργειες μακροοικονομικής υποστήριξης από πόρους της γεωργίας, αλλά βλέπουμε τώρα ξαφνικά να αναδύεται το ίδιο πρόβλημα και αυτό θα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στην συνδιαλλαγή αύριο και τις επόμενες ε, μέρες, ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ένας τρόπος που θα μας επιτρέψει να καλύπτουμε τέτοιες περιπτώσεις χωρίς να βγάζουμε χρήματα από τον προϋπολογισμό της γεωργίας. Ναι, όλα αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο χειρισμοί σε επίπεδο προπολογισμού. Γιατί αυτά τα χρήματα τη γεωργία έρχονται από τα κρατημέλη, τα κρατημέλη θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να τα βάλουν κατευθείαν στο ΙΤΕΡ. Αλλά αυτή τη στιγμή τίθεται ένα θέμα αρχή και διαχείριση του προπολογισμού. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και πάλι στο μέλλον πλεονάσματα σε ένα τομέα όπω είναι η γεωργία για να χρηματοδοτήσουμε ένα βιομηχανικό σχέδιο. Και η γεωργία και το ΙΤΕΡ παραμένουν από τι προτεραιότητε τη Επιτροπή μα. Ο James Ellis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω από τα χείλη του Γενικού Διευθυντού το πώς διαγράφεται τώρα η χρηματοδότηση δεδομένου ότι έχουμε αλλάξει τώρα τη χρηματοδότηση από το αρχικό ποσό ε, βρισκόμαστε τρεις φορές σε, σε τρεις φορές υψηλότερο επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια ενημερωμένη, επικαιροποιημένη πρόβλεψη για το πότε θα πρέπει να τελειώσει αυτή η χρηματοδότηση. Επίσης, επειδή ενδιαφέρει και την εκλογική μου περιφέρεια, θέλω να ξέρω πότε θα τελειώσει η λειτουργία του JET, που είναι το βασικό σχέδιο το οποίο εκπαιδεύει ε, επιστήμονες για το ITER, γιατί μου είπε ο διευθυντής του JET ότι μπορεί να βρεθούμε στη δημιουργία ενός συστήματος όπως το ITER, που να μην έχει αρκετό προσωπικό γιατί δεν έχουμε καταφέρει να τους εκπαιδεύσουμε πλήρως στο πρόγραμμα JET. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα γίνει για το πρόγραμμα JET και να μου πείτε αν εμείς ως Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε από τα συμβόλαια που έχουν να κάνουν με την κατασκευή Twitter και θα έχουμε αρκετή ενέργεια από την θερμοποιητική σύνδεξη. Ο Παύλου Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις στο διακρατικό επίπεδο, γιατί δεν υπάρχουν χρηματικά προβλήματα μονάχα στην Ευρώπη, αλλά και μεταξύ των εταίρων μας. <clears throat> Υπάρχει μια συμφωνία η οποία προβλέπει μια ορισμένη στάθμιση των ψήφων. Θα υπάρξει τώρα ε, μετά, θα υπάρξει τροποποίηση της ισορροπίας των ψήφων μετά από την ε, πρόταση αυτή που προτείνει η Κομισιόν και πώς ακριβώς προβλέπει η Κομισιόν να γίνουν τα πράγματα στο μέλλον. Επίσης, αν θα χρειαστεί μια νέα νομική βάση για την ε, τροποποίηση αυτή σε ό,τι αφορά την φάση της οικοδόμησης αυτού του συστήματος και επίσης τη στιγμή που βλέπουμε ότι είναι τόσο μεγάλα τα ποσά τα οποία ε, τα οποία χρησιμοποιούνται θα υπάρξει κάποια, κάποια περιορισμένη πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα περιοριστούν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος μόνο σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και management. Και το τελευταίο μου ερώτημα είναι αν μπορούμε να έχουμε ένα business plan το οποίο θα μας δείξει πώς θα μπορέσει να προχωρήσει η κατασκευή του ITER τι θα γίνει αν δεν δώσουμε τα απαραίτητα ποσά και τι θα γίνει αν περιορίσουμε τη χρηματοδότηση αυτή. Ποια θα είναι κατά ένα δισεκατομμύριο. Ποιες θα είναι οι συνέπειες των τριών αυτών σενάριων για το σχέδιο ΙΤΕΡ. Σας ευχαριστώ. Όπως πολύ ωραία είπε ο Ράιμερ Μπέρκερ, εγώ είμαι εκπρόσωπος ενός από, τα, από τις διαβόητες πολιτικές ομάδες που είναι εναντίον αυτού του σχέδιου. Και δεν είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα και η Γκουε έχει αντίθετη άποψη για αυτό το σχέδιο και υπάρχουν πολλοί από εμά οι οποίοι δεν συμφωνούν με την άποψη της πολιτικής ομάδας και τουλάχιστον έχουν εκπράξει, εκφράσει το σκεπτικισμό τους για αυτό το πρόγραμμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα αυτό το σχέδιο δεν θα είναι ποτέ επιτυχές. Όχι. Υπάρχουν ορισμένοι επιστήμονες που λένε ότι θα τα καταφέρουμε, οι άλλες πολιτικές ομάδες λένε θα τα καταφέρουμε. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο είναι στη βάση της επιχειρηματολογίας μας ως πρασίνων, το ερώτημά μας είναι κατά πόσο είναι σόφρον, κατά πόσο είναι ευφυές το να ρίξουμε τόσα πολλά λεφτά σε ένα συγκεκριμένο μοναχα σχέδιο, ενώ δεν χρηματοδοτούμε άλλα προγράμματα τα οποία μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία γνωρίζοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να είναι επιτυχή και μάλιστα σε ένα περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό πολιτικό ερώτημα, το ερώτημα της κατεύθυνσης που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και εμείς έχουμε καταλήξει σε μία άλλη άποψη από εσά. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ε, χρηματοδότησης. Η Άννη Γέντσεν τόνισε ότι υπάρχουν άλλα σχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με το περιβάλλον που λέει ότι δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Ο Σαλβαδο Γκαρίκα είπε ότι δεν μπορούμε στο Δινεκέ να παίρνουμε τα χρήματα από τη Γεωργία. Πρέπει λοιπόν να θέσετε το ερώτημα αν υπάρχει πλειοψηφία για τη χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου, να μας πείτε από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα και δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή πολιτική να λέτε ότι δεν έχουμε αρκετά λεφτά για το α πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να βρούμε για το δεύτερο, για το τρίτο πρόγραμμα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί το Συμβούλιο με τον τρόπο αυτό να αναδιανέμει τον προϋπολογισμό ο οποίο έχει καταρτιστεί από την αρχή του προϋπολογισμού και επομένω οι πράσινοι σας είπα ότι δεν υποστηρίζουν να χρηματοδοτήσουμε αυτό το σχέδιο και θέλω να ρωτήσω τον Σαλβαδόρ Γαρίγκα αν δεν πρόκειται να υπάρξει ανα διανομή των πόρων του προπολογισμού, πώς θα μπορούσατε να σκεφτείτε την φορολογία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Και φυσικά θα ήθελα να έρθω και στο θέμα της διαχείρισης. Το έχει θίξει και ο κύριος Ρούμπικ, όχι για, τελευταία, για πρώτη φορά. Ακούσαμε πολλές φορές την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα διαχείρισης. Ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε και από την Κομισιόν να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν έχουμε ένα πρόγραμμα εν εξελίξη, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα στην διαχείριση αυτού του σχεδίου είναι πραγματικά αμφισβητήσιμο για μένα αν έχει νόημα να κινητοποιήσουμε τόσο μεγάλα ποσά όσο ζητούνται σήμερα. Ευχαριστώ Χέλγα. Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν μπορεί να διαπιστώνει ότι πολλές ομάδες αλλά και πολλές διαφορετικές εθνικότητες μετά από την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία Δίνω το λόγο στον συνάδελφο για τη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για το σχέδιο Ίτερ. Αναφέρθηκαν εδώ οι διάφορες δυσκολίες και είναι πολύ καλό ε, που γίνεται διαβούλευση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στις αρμόδιες επιτροπές. Υπήρξε θέμα διάρθρωσης του σχεδίου, εύνομης διαχείρισης, υπήρχε ένα πρόβλημα διαχείρισης ε, του Ινστιτούτου της Βαρκελών και όλα αυτά βελτιώνονται. Υπάρχει, υπάρχει μια αλλαγή κατεύθυνσης λοιπόν σε αυτό το σχέδιο, έχουν ληφθεί μέτρα και ορισμένες βελτιώσεις ε, θα γίνουν ε, αρκετά σύντομα. Να θυμίσω ένα-δυο πράγματα. Καταρχήν εμείς βρισκόμαστε στα πλαίσια μιας διεθνούς συμφωσμίας που δεσμεύει την Ευρώπη ε, εναντί του υπολείπου κόσμου. Πρόκειται λοιπόν, θέλουμε δεν θέλουμε, για κάτι το οποίο δεσμεύει συνολικά τα κοινοτικά όργανα για το θέμα. Έχουμε τώρα μπροστά μας μία βιομηχανική πρόκληση μπροστά μας. Θέλουμε όντως να ορίσουμε μία νέα βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη, όπως φαίνεται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχει νόημα. Και το ΙΤΕΡ μπορεί να αποτελεί μία από αυτές τις απεικονίσεις της νέας βιομηχανικής πολιτικής. Λοιπόν, ή εμείς θα θεωρήσουμε αυτό το σχέδιο κακό, και να πούμε δεν το αρχίζουμε ή να πούμε ότι είναι καλό και το πάμε μέχρι τέλους. Δεν μπορούμε ποτέ να διακόπτουμε ένα σχέδιο στη μέση, είναι ότι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Υπάρχουν τώρα και οικονομικές προκλήσεις. Πρέπει να κάνουμε όμως μια διαφοροποίηση μεταξύ της βιομηχανικής και της οικονομικής προσέγγισης του ΙΤΕΡ. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να βλέπουμε τα πράγματα μόνο από μια οπτική γωνία. Λοιπόν, δημοσιονομικά τι λέω εγώ, ότι δύσκολα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εγώ δεν θέλω το ίτερ να λειτουργεί διορθωτικά ε, ως διορθωτικός παράγοντας άλλων οικονομικών πολιτικών. Δεν θα πρέπει εμείς να κουτσουρεύουμε άλλους, άλλες πολιτικές, ε, όπως ας πούμε η γεωργική πολιτική, για να χρηματοδοτούμε το ίτερο. Και πάμε εδώ σε ένα σημείο, το οποίο είναι ένα σημείο που αρέσει πολύ στον πρόεδρό μας, είναι το πώς θα χρηματοδοτήσουμε όχι μόνο βραχυπρόθεσμα το ίτερ, αλλά μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το πώς δηλαδή το ίτερ θα γίνει ένα μακρόπνοο σχέδιο, πώς θα του διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα έχουμε κοινοτικοποίηση ορισμένων δαπανών, θα του δώσουμε ίδιους πόρους, πώς θα βρούμε λοιπόν εμείς αυτή τη λύση για τη λύση που θα δοθεί φέτος είναι μια λύση η οποία δεν θα είναι ένα Αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική πολιτική πρόκληση για την Ευρώπη του αύριο. Έχουμε λοιπόν εμείς σε μεγάλα διαρθρωτικά σχέδια Πρόκειται για σχέδια τα οποία δεν μας έχουν πέσει από τον ουρανό, που δεν έχουν επίπτωση στους πολίτες. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς δεχόμαστε για να ε, ικανοποιήσουμε ε, την, ε, την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για ένα οικονομικό και κοινωνικό σχέδιο που χρειαζόμαστε αυτή την πρόκληση για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε όμως από την άλλη μεριά και οι ευρωπαϊκές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ελπίζω ότι θα υπάρξει πραγματικά μια στράτευση και θα μπορέσουν και πολλοί βουλευτές να πάνε στο Κανταράς επιτόπου να δούνε το σχέδιο και θα πρέπει λοιπόν εμείς να ε, μπορέσουμε να διορθώσουμε τα και κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση. Ξέρω ότι θα βγει μια ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική αυτή τη βδομάδα και αναμένω όχι μόνο να τεθεί μια σειρά από στόχους, αλλά και προτάσεις για χρηματοδότηση ώστε να ευδοκιμήσουν αυτά τα προγράμματα και σχέδια και να διατηρηθεί η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Μα γι' αυτό έχουμε εδώ το Γενικό Διευθυντή, αλλά πρέπει να το αφήσουμε και λίγο χρόνο να μπορέσει να μιλήσει. Ο Γιώραν Φέρμ έχει το λόγο, ξέρω ότι θα είναι σύντομο. Θα θέσει σωστά ερωτήματα και μετά ο Γενικό Διευθυντής, ο Γιώραν. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Δύο μονάχα σκέψει. και κάποια ερωτήματα για τη διεθνή δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Ίσως θα ήταν καλό πρώτα να εξασφαλίσουμε τη μακροχρόνια χρηματοδότηση και μετά να υπησέλθουμε σε διεθνείς δεσμεύσεις. Δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό από την αρχή. Αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση διότι μας ζουλάει η Κομισιόν μας πιέζει. Λέει ότι έχετε μια διεθνή δέσμευση και πρέπει να την τηρήσετε. Μήπως θα ήταν καλύτερο να έχουμε πρώτα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Δεύτερο ερώτημα. Η ομάδα μου δεν είναι κατά του σχεδίου ΙΤΕΡ, αλλά δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι αυτό είναι η μόνη και πρώτη προτεραιότητα στην κατηγορία 1α. Υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Φοβόμαστε ότι αυτό μπορεί να υπάρξει να είναι ακριβώς κάτι που θα οδηγήσει στην ανάγκη να περιορίσουμε άλλες δαπάνες στην κατηγορία 1α που είναι εξίσου και πιο σημαντικές. Εξίσου σημαντικές και περισσότερο. Πιστεύει η Κομισιόν ότι αυτό είναι το νούμερο 1 στην κατηγορία 1. Και είναι τόσο σημαντικό το ΙΤΕΡ που μπορούμε να περικόψουμε άλλε προτεραιότητε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή συνάδελφοι. Ο κύριο Γενικό έχει το λόγο. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Είναι ευχαρίστησή μου που βρίσκομαι εδώ για πρώτη φορά. Ορίσκα Γενικός Διευθυντής για την έρευνα. Από αύριο θα λέγεται έρευνα και καινοτομια Πρώτη 1η Ιουλίου πήρε τη θέση μου και το πρώτο θέμα που είχα στο γραφείο μου ήταν για την πρώτη Ιουλίου μέχρι σήμερα κάθε μένα ξαναγυρίζει στο γραφείο μου ο φάκελος ΙΤΕΡ. Είναι πολύπλοκο το θέμα να είναι είναι δυσκίνητα, ναι, είναι. Έχουν προβλήματα, φυσικά. έγινε λάθη, φυσικά. Μας παίρνει να σταματήσουμε τα προγράμματα ή να μην τα συνεχίσουμε. Όχι. Αν θέλετε πραγματικά να πετύχουμε τους στόχους μας για το περιβάλλον, την ενέργεια, δεν είναι δυνατόν να μην επενδύσουμε στην σύνδεξη Φερρυπίνα. Να σας δώσω ένα νούμερο ενδιαφέρον το συνολικό κόστος για το ΙΤΕΡΑ είναι 6,6 δις. Πάρα πολλά λεφτά. Αλλά είναι περίπου τα ίδια λεφτά που κάθε μέρα, κάθε μέρα ξοδεύουμε για πετρέλαιο. 6,6 δις. Πετρέλαιο βενζίνη. Ξαναγυρίζω στο κόστος και έχω και τη συνάφρα του Σαν σαν από την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών που θα μιλήσει για τα δημοσιονομικά θέματα. Αύξηση του κόστους Ξέρετε ότι το πρόγραμμα ε, σημείωσε μεγάλη αύξηση κόστους. Η συμφωνία για το ίτερ υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2006 με βάση αρχικής εκτίμησης του 2001 και η επιστημονική κοινότητα για τη σύνδεξη στα καλτιμέλη τότε το ενέκριναν. Μια από τις πρώτες δράσεις της οργάνωσης του Ίτερ από το 2007 και μετά ήταν να εκτελέσει μια αναθεώρηση του προγράμματος, του σχεδίου προγράμματος και είναι μια αναθεώρηση του κόστους. Το παρουσιάσαμε, στο, στο Συμβούλιο του Ιούνιο του 2006 πολύ πιο πάνω από το αρχικά προβλεπόμενο. Λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους η Κομισιόν ζήτησε ανεξάρτητες αξιολογήσεις αξιολόγηση κόστους να γίνει σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο και στα μέσα του 2009 όλες οι εξωτερικές αξιολογήσεις επιβεβαίωσαν την φερεγγιότητα αυτών των νέων εκτιμήσεων και ήταν σαφές ότι το πρόγραμμα αντιμετώπιζε σημαντικές αυξήσεις στο κόστος. Και γι' αυτό κάναμε προτάσεις τον Ιούλιο. Και ο συνάδελφός μου θα αναφερθεί στις προτάσεις αυτές σε λίγο. οι προτάσεις δεν είναι για να περιορίσουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Το 1 τρίτο maximum από τα κονδύλια αυτά, 1,4 πρέπει να προέρχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο. Έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν και οι άλλες προτεραιότητες στο πρόγραμμα του 2020. Ένα σωρό άλλα μέτωπα. Τώρα για τη διαχείριση. Υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Και για τη διακυβέρνηση, θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Με βάση τα ε, πορίσματα των αξιολογήσεων, η Κομισιόν πίεσε για να πετύχει να αντικατασταθούν διευθυντές της οργάνωσης και της ενέργειας σύνδεξης και να οριστούν νέοι managers οι οποίοι επελέγησαν με βάση την εμπειρία τους, τα προσόντα τους και όχι την πολιτική τους προέλευση ή την εθνικότητά τους. Οι νέοι διορισμοί μας καλύπτουν. Ο Φρέν Βίσλο, που είναι διευθυντής ε, για ενέργεια με σύνδεξη κάθε δίπλα μου, έχει διαχειριστεί τέτοιου είδους υποδομές στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Και είναι ο μόνος σωστός υποψήφιος για τη θέση αυτή, ε, για τη μονάδα που λειτουργεί στη Βαρκελόνη σύνδεξης. Η Διεθνής Οργάνωση Ίτερ είχε αντικαταστάσεις και στην διοικητική της δομή ήρθε ο καθηγητής Μοντοζήμα, νέος γενικός διευθυντής, αυτός έχει τεράστια εμπειρία, έχει κάνει παρόμοιες εγκαταστάσεις στη χώρα του ήδη. Οπότε η οργάνωση είναι έτοιμη για το στόχο της. Και δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και η υποδομή. Θέλουμε να βελτιωθεί το management, η οργάνωση, η εσωτερική έλεγχη και ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να μην έχουμε νέες υπερβάσεις κόστους και με σωστό management. Τις επόμενες εβδομάδες θα σας υποβάλουμε και στα κράτη-μέλη μία ανακοίνωση για το πώς τα μέτρα αυτά του management, της διαχείρισης, αριστοποίησης του management και μείωσης του κόστους, πώς θα εφαρμοστούν. Ο Φραν Μπίσκο που κάθεται δίπλα μου ήδη εισήγαγε τα, το πρώτο από τα μέτρα αυτά έστω ότι το πρόγραμμα να μπορεί να κινηθεί με βάση το ε, χρονοδιάγραμμα που έχει επιλεγεί για τη διακυβέρνηση governance στην ανακοίνωση που θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες θα δείτε συγκεκριμένες ιδέες για να βελτιωθεί ο ρόλος της Ένωσης. Γιατί στην δομή διακυβέρνηση δεν έχουμε το μερίδιο που δικαιούμαστε. Αυτό δεν μας επιτρέπει να παίξουμε το ρόλο που θέλαμε να παίξουμε σε αυτή την οργάνωση. Θα δείτε συγκεκριμένες προτάσεις στις επόμενες εβδομάδες. Τέλος για το JET, το Joint, Undertaking που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και που είναι προκειμένου να προωθηθεί, να προχωρήσει το πρόγραμμα ITER. Αυτή η οργάνωση ήδη ενισχύεται και θα εξακολουθεί να ενισχύεται από κοινωνικά κονδύλια. Φτάνει το τέλος της ζωής της γύρω στη 2015, τουλάχιστον αυτό λένε οι πυρογνώμονες και πρέπει η γνώση να μεταφερθεί από το Jetty Column στο ITER και το προσωπικό επίσης σιγά σιγά να μεταφερθεί. Μοναδική εμπειρία είναι αυτή στην Ευρώπη και χρειάζεται προκειμένου να προοδηθούν τα προγράμματα αυτά. Εγώ λοιπόν είμαι αισιόδοξο με τη νέα δομή του management. Με τις ιδέες που θα δείτε για τη συγκράτηση του κόστους θα μείνει το πρόγραμμα μέσα στο ρυθμό του χρονοδιαγράμματος και το πρόγραμμα είτε επαναλαμβάνω, θα κρατηθεί μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος. Επιτρέψτε κύριε Πρόεδρε, ο συνεργάτης μου να αναφερθεί στο δημοσιονομικό σκέλος της πρότασης. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Διευθυντά. Ο Γενικός Διευθυντής του Προπολογισμού θα γίνει να προσθέσει κάτι. πολύ σύντομα, γιατί νομίζω θα αναφερθεί το θέμα αύριο αυτό στη συνδιαλλαγή. Ο συνάδελφος σας εξήγησε από πού ερχόμαστε, τι προβλήματα συναντήσαμε και όλοι ξέρουμε τις συνθήκες κατά τις οποίες μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις ανάγκες. Ακούσαμε το μήνυμα του Κοινοβουλίου που ζητάει μια πιο πλήρη εικόνα της μεθόδου χρηματοδότησης. Αύριο θα προσπαθήσουμε να σας διαφωτίσουμε όσο γίνεται. Δεν νομίζω έχει νόημα τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει το θέμα το θέμα της χρηματοδότησης από το κεφάλαιο 2 είναι γνωστό 11 μέρες πριν τελειώσει η γεωργική καμπάνια για το έτος 2010 μας επιτρέπει να είμαστε καλά πληροφορημένοι και χωρίς λάθος για τα ποσά που είναι διαθέσιμα στο κεφάλαιο αυτό αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα ποσά που προβλέπτηκαν προβλέφτηκαν για το 2010. Αν δεν γίνουν μεταφορέ, θα χαθούν τα χρήματα αυτά και τότε θα έχουμε πραγματικό πρόβλημα χρηματοδότησης Twitter. Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρίσκο που είναι διευθυντής της ενέργειας σύνδεξης είναι εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που είπε ο Γενικός Διευθυντής. Σα Σας ευχαριστώ. Ίσως μπορώ να κάνω μια σύντομη δήλωση σχετικά. Να σας πω ότι φυσικά το ITER είναι ένα μεγάλο επιστημονικό εγχείρημα, αλλά ιδίω αυτά τα δέκα χρόνια απετέλεσε και ένα τεράστιο κατασκευαστικό σχέδιο. Όταν ξεκίνησα, <clears throat> όταν ανέλαβα τις ε, το αξίωμα αυτό στην Βαρκελόνη το 2010, το Φεβρουάριο. Κατάλαβα ότι χρειαζόμαστε καλύτερη διαχείριση σχεδίου από το ίτερ. Είχαμε πολύ καλή ομάδα για τα τεχνικά θέματα, για τις συμβάσει, αλλά δεν είχαμε αρκετή ικανότητα σε επίπεδο διαχείρισης σχεδίων, project management. Έχω λοιπόν δώσει έμφαση σε αυτόν τον τομέα τους πρώτους αυτούς μήνες. Έχω μια σειρά από προτάσεις για να τροποποιηθεί η οργανωτική δομή του ΙΤΕΡ για να είναι η διαχείριση των σχεδίων το κέντρο της εργασίας μας. Θα υπάρξει και αλλαγή σε επίπεδο προσώπων μέσα στη δομική αλλαγή. Και επίσης θέλω να αλλάξω ορισμένε διαργασίες που χρησιμοποιούμε σε επίπεδο διαχείρισης, χρησιμοποιώντας τις φυσιολογικές πρακτικές οποιοδήποτε βιομηχανικού σχεδίου τέτοιας κλίμακος και είναι πρόθεση μου να τροποποιηθεί το σύστημα αναφορών, ώστε τόσο εκθέσεων και αναφορών, ώστε τόσο εσωτερικά όσο και προς τον έξω κόσμο, θα είναι σαφέστερη η πρόοδος στο έργο μας. Έχω κάνει λοιπόν αυτές τις προτάσεις. Ήδη εδώ και κάποιους μήνες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και στις 5 Οκτωβρίου ανεκρίθησαν. Έχω κάνει τις πρώτες αλλαγές στην δομή και αυτή τη βδομάδα είχα συναντήσεις με τους, πρώτους, με τους νέους ηγέτες των ομάδων project που είναι στο κέντρο της νέας δομής και απλώς θέλω να πω ότι όχι μονάχα συζητούμε τις αλλαγές αλλά οι αλλαγές αυτές γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Για την συγκράτηση του κόστους. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα με την διαχείριση σχεδίων, είναι ένα κομμάτι της διαχείρισης σχεδίων, <clears throat> αλλά επιπλέον μπορώ να σας διαβεβαιώσω λιγάκι για την συγκράτηση του κόστους. Τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν προέρχονται από επισκοπήσεις πριν από δύο ή τρία χρόνια και όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής είχαν επικυρωθεί από ανεξάρτητους ελεκτές. Αλλά δεν υπήρξαν και είμαι ευτυχής γι' αυτό δυσάρεστες εκπλήξεις τον τελευταίο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο δεν νομίζω να έχουμε ανακαλύψει κάτι συγκεκριμένο αρνητικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του κόστου Twitter. Και ορισμένα από τα μεγάλα <clears throat> συμβόλαια, κάποιες από τις μεγάλες συμβάσεις για την κατασκευή του Twitter έχουν ήδη συναυθεί και η εμπειρία μας είναι ότι οι τιμές τις οποίες, στις οποίες γίνονται οι συμβάσεις αυτές είναι χαμηλότερες από τις αρχικές μας προβλέψεις. Ώστε με όλα αυτά νιώθω μεγαλύτερη άνεση με τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν προβλέπονται άλλες αυξήσεις κόστους για το ΙΤΕΡ. Επιπλέον αυτό το σχέδιο πια είναι πολύ πιο προχωρημένο. Όταν έγιναν οι πρώτες εκτιμήσεις κόστους πριν από 2-3 χρόνια ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού δεν είχε ακόμα συμπληρωθεί και υπήρχαν πολλά χάσματα και κενά. Αλλά τώρα έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Πολύ, ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού είναι, έχει και ξεκινάει τώρα η κατασκευή. Στην Κανταράσου θα δείτε λοιπόν τα πρώτα κτίρια τα οποία εμφανίζονται στην πλατφόρμα η οποία είχε δημιουργηθεί για αυτόν τον στόχο και σε διάφορα σημεία της Ευρώπης γίνεται η κατασκευή μερικών από τα κύρια συστατικά στοιχεία του αντιδραστήρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Κύριε Σιγητά, θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Όπως είπε και ο Γενικός ε, Διευθυντής, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα αύριο στην συνδιαλλαγή και τον τριγωνικό διάλογο. Δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία είπαμε θα πρέπει να ερμηνευθούν ως δυσπιστία προς εσάς. Αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ ε, ενθαρρυντικά, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα καθόλου ποιες θα είναι οι οριστικές προτάσεις για το management του σχεδίου αυτού και κατά πόσο θα τύχουν έγκρισης και θα μπορέσουν πράγματι να εφαρμοστούν. Αν αν έχουμε μια συμφωνία στις 11 Νοεμβρίου στο τέλος της ε, διαδικασίας ε, αυτής θα μπορούσε να υπάρχει η απόφαση για περαιτέρω χρηματοδότηση. Δεν ξέρω λοιπόν γιατί γιατί δεν μπορούμε να δεν κατάλαβα αυτό που είπατε για, τις αγροτικές, για τους αγροτικούς πόρους του 2010, ότι θα χαθούν αν δεν βρούμε κάποια συμφωνία. Με. Συγγνώμη, αυτοί οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς άλλους τρόπους. Μπορούμε με ένα διορθωτικό προϋπολογισμό να κάνουμε πολύ πιο σημαντικές αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Ξέρουμε όμως ότι στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και κοιτάζω τον ε, Παύλου Ρέμπιχ και ξέρουμε ποιες είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Αυστρίας, η μεταρρύθμιση που προτείνεται από την Κομισιόν απορρίπτεται από την Αυστρία. Δεν γνωρίζω αν μόνο μια χώρα η οποία θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, να απορρίψει και να μην δεχτεί μια τέτοια μεταφορά αυτών των ποσών σε άλλη κατηγορία. Απλώς θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ήταν οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι έλεγξαν τα στοιχεία αυτά που μας έφεραν σε μια απόφαση η οποία σήμερα μας αναγκάζει να ζητούμε πρόσθετη χρηματοδότηση 1,4 δισεκατομμύρια. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουμε και πάλι αυτά τα ποσά, ότι δεν θα έχουμε μια δυσάρεστη έκπληξη στο μέλλον αφού θα έχουμε ήδη κάνει τις προβλέψεις μας σε επίπεδο δημοσιονομικών προοπτικών και θα ήθελα επίσης να γνωρίζω τι σημαίνει αυτό το οποίο λέτε για τις 12 Οκτωβρίου όπου ο Γενικός Διευθυντής είχε πει ότι με το τέλος του χρόνου θα λάβει η χώρα μια δημόσια ακρόαση για αυτό το σχέδιο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση, και τι θα περιλάβει και αν αυτή η δημόσια κρόση θα τροποποιήσει και το, το κόστος του σχεδίου. Επίσης για το χρονικό ορίζοντα η Κομισιόν μπορεί να μεταφέρει χρήματα από το 2010 στα έτη 2011 έως 2013 Επομένως, η χρηματοδότηση δεν θα αφορά το 2010, αλλά το 2012 και το 2013. Επομένως, αυτή τη στιγμή βέβαια τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει αυτό με οποιοδήποτε τίμημα και κυρίως με το να παραμελήσουμε άλλες ε, δραστηριότητες στον ερευνητικό τομέα που είναι και αυτό προς το δικό σας συμφέρον, γιατί πολλές από αυτές τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ερευνητικό επίπεδο θα είναι χρήσιμες και για το δικό σας σχέδιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούμε σε ένα σόφρον επίπεδο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα εγγυάται ότι αυτό το οποίο εσείς παρουσιάσατε ως πρόταση να μπορεί να ενταχθεί με ένα πιο επακριβή τρόπο στις δημοσιονομικές προοπτικές. Εγώ λέω τώρα, χωρίς να σκεφτώ ιδιαίτερα, χωρίς να έχω προετοιμάσει κάτι. Ας πούμε ότι βρίσκουμε μια λύση για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το ΙΤΕΡ χωρίς να θίξουμε τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάξει, αλλά τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι άλλες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν, θα ληφθούν για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε όλα αυτά τα ποσά τα οποία είναι απαραίτητα για το ΙΤΕΡ. Και φυσικά και η δική μας πρόταση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πρόταση την οποία θα μας υποβάλει η Κομισιόν στην αρχή του τρίτου μέρους διαλόγου και της συνδιαλλαγής που θα ακολουθήσουμε το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά, σας άκουσε η Κομισιόν. Κατά τον τελευταίο δημοσιονομικό τρίλογο συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο να οργανώσουμε στην αρχή της επόμενης χρονιάς μία κοινή αποστολή επιτόπου. Ασυνήθιστο αυτό. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και φυσικά και Κομισιόν θα έρθει. Επιτόπου. Προς στιγμήν είπαμε Κανταράσο. Αλλά τα πιο σημαντικά όμως ε, διαμείβονται στη Βαρκελόνη. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε και στο γιαπί και στο χώρο από όπου γίνεται η διαχείριση όλου του σχεδίου. Όπως ανέφερε ο εισηγητής μας, οι προτάσεις που έθεσε η Κομισιόν για να αρχίσει να χρηματοδοτεί την επιπλέον χρηματοδότηση που χρειάζεται δεν έχει λυθεί ακόμη για την περίοδο 2010-2013. Με όλη αυτή δηλαδή την επικίνδυνη ακροβασία όπου εμείς ε, παίρνουμε τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα το 2010 και αρχίζουμε να τα ξοδεύουμε το 2012, το πρόβλημα θα τεθεί το 2013. Οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, υπό την ε, αρμοδιότητά σας κύριε Γενικέ, ελπίζουμε ότι θα δώσουν τα προεξοφλημένα αποτελέσματα. Αλλά όπως είπανε, δεν αφισβητούμε την εξουσία, αλλά όπως είπαν οι συνάδελφοι, είναι ένα σχέδιο πάρα πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να αποφύγει. Αλλά οι οικονομικοί μας, οι οικονομικές μας δεσμεύσεις είναι τόσο σημαντικές και είμαστε τόσο σφιγμένοι οικονομικά που πρέπει να βρούμε μια λύση. Λύνουμε, τελειώνουμε λοιπόν τη συζήτηση σε αυτό το σημείο. Υπενθυμίζω ότι θα κρατήσουν, θα μείνουν εδώ οι συντονιστές για μια ώρα. Και η επόμενη συνεδρίαση των, της Επιτροπής Προπολογισμών θα γίνει 9 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Θα αρχίσουμε δηλαδή 9 το πρωί μέχρι τις 6.30. Δηλαδή, ευχαριστώ πέρα στη συνεδρίαση.